Καλή σας μέρα. Ε, προσπάθησα να καθυστερήσω ελπίζοντας ότι θα έρθουν διάφοροι κι άλλοι στην Επιτροπή μας. Εν πάση περιπτώσει, ε, εγκρίνεται την ημερήσια διάταξη τι θεωρώ εγκεκριμένη. Τώρα, ανακοινώσει του Προέδρου δεν υπάρχουν. Πάμε κατευθείαν στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιδιωτικά συστήματα». Ο κύριος Κούτας είναι ο εισηγητής. Βεβαίως υπήρξε εδώ σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Εμείς φτιάχνουμε γνωμοδότηση γιατί θεωρήθηκε ε, από την συνδιάσκεψη των Προέδρων ότι επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή Απασχόλησης. Τέλος πάντων, για τα σημεία 2, 5, 10, 11 και 12 έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα εμείς, αλλά για τα σημεία 6, 7, 9 και 14 έχουμε, έχει την αρμοδιότητα η Επιτροπή Απασχόλησης. Ή ε, έχουμε, συγγνώμη, κοινή αρμοδιότητα με την Επιτροπή Απασχόλησης. Η Επιτροπή Απασχόλησης βεβαίως ε, είπε ότι αν κατατεθούν τροπολογίες ε, για θέματα που είναι της άμεσης αρμοδιότητας Επιτροπής Απασχόλησης θα απορριφθούν ε, εξ αρχής. Δεν θα γίνουν αποδεκτές. δεν ξέρω, εμείς αναφέραμε την... τις αντιρρήσεις μας τέλος πάντων. Μπάς περιπτώσει αν έχετε τροπολογίες αποφασίστε τι θα κάνετε. Έχετε το λόγο κύριε Κουτάς. Ναι. Ελπίζω, κυρία Πρόεδρε, αυτό που μόλις τώρα περιγράψατε να μην συμβεί. Συζήτησα με τον εισηγητή, με την εισηγήτρια από την Επιτροπή Απασχόλησης και υποσχέθηκε ότι θα έχουμε καλή συνεργασία και τελικά δεν θα απορριφθούν τροπολογίες μας ακόμη και να αφορούν θέματα δικής τους αρμοδιότητας. Τέλος πάντων, για την έκθεση αυτή αυτή κάθε ε, λέμε ότι επουδενή λόγο μπορούμε να φανταστούμε ενιαία ομοιόμορφα συνταξιοδοτικά συστήματα. Είναι εθνικά τα συστήματα αυτά και υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Ε, α, από εκεί και πέρα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο παραδείγματος χάρη για την ευελιξία, στην εργασία, για κανόνες φερεγγιότητας, για χίλια δυο πράγματα. Επίσης έχουμε ένα κάποιο υπάρχει ήδη ένα κάποιο πλαίσιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συντάξεις ε, και λέγεται ότι πρέπει να ε, υπάρχει επάρκεια βιωσιμότητα και ασφάλεια στα σταξιοδοτικά συστήματα ε, από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν ε, διαφορές όπως είπαμε και τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να τροποποιήσουν, να προσαρμόσουν τα συνταξιοδοτικά του συστήματα. Και επειδή πραγματικά εδώ πρόκειται και ε, ουσιαστικά για ένα εργαλείο soft law, ε, πραγματικά ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ε, ανταλλαγή και υιοθέτηση αν θέλετε των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών το σύμφωνο σταθερότητας επίσης αναφέρεται ε, σε ορισμένα θέματα που σχετίζονται με τα που θα μπορούσε να πει κανείς ότι συνδέονται με τα ε, συνταξιοδοτικά συστήματα γιατί τη για προστασία των ασφαλιστικών συστημάτων κτλ. Μιλ, Βεβαίω, από εκεί και πέρα η σταθερότητα ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν μπορεί να είναι ξένη προς, την, προς τα συνταξιοδοτικά ε, συστήματα που, που εφαρμόζονται. Από εκεί και πέρα η οποιαδήποτε μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων κοστίζει και ε, ε, αυτό και στην πράσινη βίβλο πραγματικά αναφέρονται οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εν ώψη αυτών των προσαρμογών. Ε, αναφέρεται η γύρενους του ευρωπαϊκού πληθυσμού όπου ε, κάποια στιγμή το, ε, ένας από τους τρεις ε, Ευρωπαίους θα είναι άνω των 60 ετών. Είναι λοιπόν πρωταρχική σημασία να ε, να προσαρμόσουμε τα εξοδοτικά συστήματα και να ανέβρουμε διαφορετικές λύσεις πηγές μάλλον χρηματοδότησης των συστημάτων τα συστημάτων αυτών ίσως θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στις εισφορές επίσης στις εισφορές από την άλλη μεριά θα πρέπει βεβαίως επειδή ε, να εξασφαλίσουμε ότι οποιασδήποτε εισφορές και δομή του σταξιοδοτικού συστήματος μπορεί να γίνουν ανεκτές από την κοινωνία και και σίγουρα τα στεξιοδοτικά συστήματα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζονται και να ισχύουν για όλους. Επαρκή βιώσιμη σύνταξη για όλους θέλουμε. Ε, ένα σύστημα το οποίο α, ε, μπορεί να το θεωρούμε εμείς βιώσιμο αλλά το οποίο προβλέπει πολύ χαμηλές συντάξεις δεν μπορεί να επιζήσει και να θεωρηθεί ικανοποιητικό. Ε, Πρέπει λοιπόν να καθίσουμε να σκεφτούμε αλλαγές. Συγχρόνως, επειδή υπάρχει και ο δημογραφικός παράγοντας και το προσδόκιμο ζωής, θα πρέπει να σκεφτούμε ε, την συνάρτηση των συντάξεων ε, από από τις παραμέτρους αυτές αλλά πριν να πούμε στον κόσμο να μένει μέχρι τα βαθιά γεράματα και να εργάζεται, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι νέοι χρειάζονται δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να εξισορροπηθούν όλες αυτές οι παράμετροι. Ε, την σήμερα ημέρα και σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν συνταξιοδοτικά συστήματα τα οποία να χρηματοδοτούν 100% από το δημόσιο. Θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αν θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να επιβιώσει. Επίσης πιστεύω ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι απλά ευάλωτοι, είναι και ε, ουσιαστικά μια κατηγορία πολιτών που είναι όμοιροι ουσιαστικά των διαφόρων κυβερνήσεων γιατί οι διάφορες κυβερνήσεις το πρώτο που κάνουν όταν υπάρχουν ελλείμματα ε, είναι ότι προσφεύγουν στους συνταξιούχους και κόβουν τις συντάξεις τους. Λοιπόν, ε, τα συντοξιοδοτικά συστήματα θα πρέπει να φροντίζουμε να δρούν σαν αναδιανεμητικά συστήματα όχι μόνο μεταξύ των γενεών αλλά μεταξύ και των ομάδων της ίδιας γενεάς. Τα συστήματα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το δημόσιο βεβαίως είναι ναι, τεράστια σημασίας και αλλά όλα τα συνταξιοδοτικά συστήματα όπως και να χρηματοδοτούνται θα πρέπει να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να υπάρχουν συμπληρωματικά συστήματα αν θέλετε τα οποία να συμπληρώνουν τα εισοδήματα από τα, αποκλειστικά δημόσια στα συστήματα. Εμείς πιστεύουμε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε μόνο με μια προσέγγιση πολλών πυλώνων και πολλών τομέων δημόσιου και μη να εξασφαλίσουμε επαρκή βιώσιμα και ασφαλή συνταξιοδοτικά συστήματα. Στη... Γι' αυτό πιστεύω ότι η αρχή για τις ευρωπαϊκές ε, επαγγελματικές για τις ευρωπαϊκές συντάξεις πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και να καθοδηγήσει τα συνταξιοδοτικά συστήματα όλων των χωρών. Τέλος να πω ότι Ε, πρακτικά δηλαδή για τη γνωμοδότηση θα έχουμε καλή συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης αλλά για να μπορούμε να έχουμε και καλά αποτελέσματα θα πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά αν θέλετε και θα ήθελα να ευχαριστήσω κλείνοντας ιδιαίτερα τον Άιβορ για την ε, συμμετοχή του και τη βοήθεια που μου προσέφερε και είμαι στη διάθεση των συναδέλφων για να ακούσω τις ιδέες τους, τις απόψεις τους. Πρόεδρος, Ευχαριστώ. Χαίρομαι που είπατε ότι έχετε καλή σχέση με την εισηγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης. Ε, αυτό πάντως το οποίο είπα εγώ για τις τροπολογίες ε, ήταν κάτι που ελέγχθη από τον πρόεδρο και ο πρόεδρος είναι αυτός που αποφασίζει για τις τροπολογίες. Η συγκήτρια μπορεί να έχει άλλη άποψη αλλά τώρα υπάρχουν σκιώδεις εισηγητές εδώ. Ωραία. Right, so maybe Danuta, you're first, because your first on my list. That makes life easier for me. Okay. Παρακαλώ. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι κατά πόσο υπάρχει επάρκεια mm, e, στην πράσινη βίβλο αυτό που έχει σημασία είναι τα συστήματα συνταξιοδότησης και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε την χρηματοπιστωτική κρίση, πώς εξελίσσεται το υπερβολικό δημόσιο χρέος καθώς και τα ε, ελλείμματα και να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια αλληλεγγύη στην Ευρώπη υπέρ των μελλοντικών γενεών. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη η νέα χρηματοοικονομική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τους συστημικούς κινδύνους και να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφασίζοντας για τη μελλοντική μορφή των συστημάτων ε, συνταξιοδότησης. Ο εισηγητής ε, το τόνισε αυτό, ότι δηλαδή ε, τα συνταξιοδοτικά βρίσκονται είναι υπό την αρμοδιότητα των κρατών μελών και τα συστήματα συνταξιοδότηση είναι πολύ διαφορετικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, άρα είναι δύσκολο να συγκριθούν. Θα ήθελα λοιπόν να λάβουμε υπόψη την επιστολή ε, που υπογράφηκε από εννέα χώρες, Ρουμανία, Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία και άλλες, που θα υπομισθούν πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος από την ε, μεταρρύθμιση αυτή και πώς θα αντιμετωπίσουμε το δημόσιο χρέος και το δημόσιο έλλειμμα. Και αυτές οι χώρες πλήττονται ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια του συστήματος ε, χρημα, ε, χρηματοδότησης του συστήματος και είναι δύσκολο να λειτουργήσουν μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Τώρα, αν κοιτάξουμε τα, τις λεπτομέρειες της έκθεσης, θα ήθελα να τονίσω ότι ο εισηγητής ε, αναφέρει ότι τα συστήματα συνταξιοδότησης θα πρέπει να οδηγούν σε ένα επαρκές εισόδημα για τους πολίτες και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα συστήματα χρηματοδότησης των συστημάτων δεν είναι τα ίδια. Διαφέρουν. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε ένα επαρκέ σύστημα συνταξιοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. Αν δούμε λοιπόν τους στόχους των συνταξιοδοτικών συστημάτων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι για να διασφαλίσουμε επαρκές σύστημα, ένα επαρκές σύστημα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ηλικία συνταξιοδότησης. Και αυτό το αναφέρει ο εισηγητής. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στην παρούσα ε, ηλικία συνταξιοδότησης και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την πρόορη συνταξιοδότηση. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν μία προτεραιότητα. Και αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε ένα επαρκές ε, σύστημα χρηματοδότησης έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτά τα συστήματα. Ως προς τα trust funds θα πρέπει να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε μέσα στα πλαίσια της μεταφοράς. Υπάρχει ανασφάλεια δικαίου σε ορισμένα ε, ως προσωρισμένα θέματα και θα πρέπει να εποπτεύσουμε την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη-μέλη και θα πρέπει να ορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να ερμηνεύσουν σωστά την οδηγία. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε ενδεχομένως και την οδηγία σε σχέση με την φερεγγιότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων και την αφαιρεγγιότητα των εργοδοτών, αυτά τα θέματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν όχι μόνο ε, δυνάμει του συστήματος Solvency 2, φερεγγιότητα 2 αυτού του συστήματος το οποίο θα εισαχθεί μετά το 2012 και δεν ξέρουμε πώς το σύστημα θα λειτουργήσει, θα πρέπει να το εντάξουμε στα πλαίσια της ε, νέας Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής που θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει το πρόγραμμα Solvency 2, οι κανόνες αυτοί, να αφορούν τα συνταξιοδοτικά ταμεία των εργαζομένων, διότι υπάρχει ιδιαιτερότητα ως προς τη, το τα συνταξιοδότηση Ορισμένοι εμπειρογνώμονε θεωρούν ότι θα πρέπει να έχουμε διαφορετικά συστήματα φερεγγιότητας και θεωρούν το πρόγραμμα Solvency 2 που θα εφαρμοστεί στα συνταξιοδοτικά ταμεία θα πρέπει να, να τύχει μίας, ε, μίας μελέτης ε, επιπτώσεων αντικτύπων πριν εφαρμοστεί αντικτύπου. δεν ähm, äh, ο συνάδελφος μου Dirk Στέρτ ε, βρίσκεται σε επαγγελματικό ταξίδι στο Μεξικό και με, παρακάλεσε να παρουσιάσω εγώ τις απόψεις του για το θέμα αυτό. Ελπίζω να μπορέσω να το κάνω σύμφωνα με το πνεύμα του Dirk. Συμφωνούμε όλοι ότι το θέμα των κανόνων των συνταξιοδοτικών συστημάτων ε, είναι το κύριο, το ο, μεγάλο αν θέλετε καυτό κοινωνικό θέμα την σήμερον ημέρα. Δεν υπάρχει καμιά μέρα, καμιά χώρα με συγχωρείτε που να μην προσπαθεί να προσαρμόσει τα συνταξιοδοτικά της συστήματα ζητήματα ε, στις παρούσες συνθήκες. Οπότε ε, δεν ε, έχει κανείς αντίρρηση για τις αλλαγές και τις αναποσαρμόσεις των δεξιοδοτικών συστημάτων συγχρόνως όμως οι χρηματοδοτικοί πόροι γίνονται όλο και μικρότεροι και τα, μ, η ανάγκη λιτότητας μεγαλύτερη γι' αυτό ο λέει ότι υπάρχουν τρία πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αν, θέλει, αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμο εξοδοτικό σύστημα. Πρώτο, πρέπει να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη η Επιτροπή μας εδώ και κάμποσο καιρό κατά κύριο λόγο ασχολείται όλο και περισσότερο με ε, νομοθετικές πράξεις για την α, ε, επιβολή κανόνων στην ε, χρηματοπιστωτική αγορά, στις αγορές γενικώ. είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να δούμε κατά πόσον μπορούμε να Δηλαδή, κατά πόσο οι αλλαγές αυτές που κάνουμε περιορίζουν αν θέλετε την, το ενδεχόμενο ανάπτυξης μήπως δηλαδή κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν αφήνουν την ανάπτυξη να ε, προχωρήσει του ρυθμούς που θα μπορούσε να ε, προχωρήσει. Οικονομική ανάπτυξη λοιπόν πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα ε, το όριο, το στε, όριο σύνταξης ε, δημογραφικοί παράγοντες, ε, προσδόκιμο ζωής και τα λοιπά επηρεάζουν τα α, όρια ηλικία. Όμως ε, ό,τι και να κάνουμε εμεί οι υπόλοιποι, τα πάμε στα 60, 62, 65 κτλ. Οι Σουηδοί μας κοροϊδεύουν γιατί αυτοί βρίσκονται ήδη στα 67 και από εκεί και πέρα προβλέπουν να αυξήσουν ακόμη τα όρια. Τέλος πάντων, τα όρια ηλικία είναι σημαντικό, σημαντική παράμετρος πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε, όπως είπε και η η προηγούμενη ομιλήτρια ε, να δούμε πώς υπολογίζονται οι υποχρεώσεις ε, των πολιτών και άρα οι εισφορές και βεβαίως τι απορρέει για τη χρηματοδότηση από αυτό. Αυτή τη στιγμή ε, στις περισσότερες χώρες η χρηματοδότηση είναι εν πολλής κρατική. Στην Γερμανία τα αποθεματικά ε, για το, στο τομέα των τη συντάξεων έχουν ένα κάποιο μέγεθος όμως δεν ξέρουμε πως θα επαρκέσουν ε, θα πρέπει όμως ε, χρόνος να σκεφτούμε ε, θέλουμε ε, πράγματι να δουλέψει τέλεια και πλήρως η κοινή εσωτερική αγορά και να προχωρήσουμε και σε μια κοινή αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είπε και ο Μάριο Μόντι αυτό. Ε, το έθεσε και αυτός αυτό το ερώτημα. Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μέχρι τώρα είχε πάρει μια κάποια θέση η οποία δεν ε, ουσιαστικά ε, ε, έλεγε ότι είναι για αργότερα και δεν συζητούμε ακόμη το κατά πόσον ένα επάγγελμα ή η δουλειά που έχει κάποιος είναι φορητή άρα μπορεί να μεταφερθεί ε, από το ένα μέρος στο άλλο ή όχι. Αλλά αν θέλουμε μια κοινή αγορά εργασίας πραγματικά θα πρέπει να αλλάξουμε θέση. Το επόμενο θέμα είναι ότι ε, οι περισσότερες χώρες έχουν τρεις πυλώνες την ε, δημόσια σύνταξη, την ε, προαιρετική σύνταξη την επαγγελματική αν θέλετε και τελικά την συμπληρωματική, επικουρική αν μπορούμε να την πούμε έτσι. Βεβαίως δεν είναι συγκρίσιμα τα συστήματα τα οποία υπάρχουν και ε, αλλά αν θέλουμε να φτάσουμε έστω και σε μία ελάχιστη εναρμόνιση εμείς εδώ στην Ευρώπη κάποια πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν από τους προηγούμενους ομιλητές ετέθησαν και άλλα θέματα τι θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή με το <laughs> τι θα κάνουμε το Solvency 1, Solvency 2 γιατί στο Solvency 1 υπήρχε μια κάποια συγκρισιμότητα αυτά τα ερωτήματα είναι θεμητά δεν είναι φήμη ούτε υποψία κάποιων. Αν θέλουμε πραγματικά να ισχύουν αυστηροί κανόνες για τη το ασφαλιστικό επικουρικό κομμάτι της σύνταξης ε, αντίστοιχα πράγματα θα πρέπει να ισχύουν και για τους άλλους πυλώνες και το, αυτό κοστίζει χρήματα θέλουμε να ακριβίνουν αν θέλετε οι, οι, οι άλλες συνιστώσεις της τελικής σύνταξης. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε κάτι τέτοιο. Είναι ένα σοβαρό ερώτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, του χάρη, που συμβάλλουν στην επαγγελματική σύνταξη, στον επαγγελματικό πυλώνα, αν θέλετε. Το Πρόβλημα βεβαίως δεν είναι κατά πόσον εμείς θεωρούμε κάτι τέτοιο εφικτό για το μέλλον. Ε, το θέμα είναι πώς θα κάνουμε τις αλλαγές αυτές και κατά πόσον θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι αλλαγές αυτές. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα μπορούσε κάλλιστα να βρει μια πρακτική ε, συμβιβαστική λύση και γι' αυτό θα θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει και μία μελέτη οικονομικού αντικτύπου. Αυτές είναι οι σκέψεις λοιπόν του συναδέλφου μου Dirk Sterks. Α, στο τέλος αναφέρεται και στο θέμα της ενημέρωσης και τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν κατανοητές πληροφορίες οι οποίες να δίνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους διότι δίχως κατανοητές και πλήρεις πληροφορίες δεν μπορεί κανείς να κάνει επιλογές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Σίγουρα και ο εισηγητής ε, θα τα λάβει υπόψη αυτά και στην Επιτροπή Απασχόλησης θα συζητηθούν φαντάζομαι όλες αυτές οι παράμετροι. Το κατά πόσο θα φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα δεν το ξέρω, διότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα, αλλά είναι και πάρα πολύ περίπλοκο. Ευχαριστώ, συμφωνώ με όσα ελέγχθησαν και ίσως θέσω τα ζητήματα κάπως διαφορετικά. Βλέπω δύο ζητήματα εδώ και ενδεχομένως τρία. Το πρώτο και που είναι θετικό είναι ότι υπάρχει υψηλότερο προσδόκιμο επιβίωσης, όλοι ζούμε περισσότερο. Όλοι μιλάμε για δημογραφικές ε, προκλήσεις χωρίς να σκεφτόμαστε τα ευεργετήματα. Και 65 ήταν ένα όριο το οποίο είχε θέσει ο Βίσμαρκ όταν οι άνθρωποι ζούσαν λίγο περισσότερο μόνο από τα 65. Εν πάση περιπτώσει, ως προς το ερώτημα της Επιτροπής, ε, πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα υψηλότερο όριο συνταξιοδότησης, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε κατά διαφορετικούς τρόπους. Είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα, αλλά δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε αυτές τις εργασίες προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλάμε για επανακατάρτιση και γνωρίζουμε ότι η εργασία που είχαμε στα 25 μπορεί να μην είναι η ίδια με αυτή των 65. Το δεύτερο ζήτημα είναι η εμπιστοσύνη στα αποταμιευτικά συστήματα. Σε, σε μια πρόσφατη ε, ε, ενημέρωση για το θέμα της αποταμίευσης είναι ότι όσο νωρίτερα αποταμιεύουμε, τόσο περισσότερα χρήματα θα έχουμε για τα γυρατιά μας. Ξέρουμε τι συνέβη στην ε, χρηματοπιστωτική αγορά και βεβαίως η επόμενη γενιά δεν θα έχει και τόση εμπιστοσύνη στο αποταμιευτικό μετά από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Το θέμα της μεταβιβασιμότητας του συνταξιοδοτικού είναι επίσης ε, σημαντικό μέσα στα πλαίσια της κινητικότητας η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν ε, μεγαλύτερη, μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με αυτό το θέμα του pension gap. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εικόνα που θα έχουμε στο μέλλον. Δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ε, μέσα, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ε, είναι ευεργετικά αυτά τα συστήματα σε σχέση με το pension gap και αυτό μας ενδιαφέρει είναι η φερεγγιότητα, το σύστημα φερεγγιότητας στη στιγμή που αποταμιεύουμε σήμερα. Μιλήσαμε για το, ε, ε, για το θέμα των συνταξιοδοτικών ταμείων, ο Πίτερ θα μας πει περισσότερα. Θα πρέπει να γίνει όμως μια μελέτη αντικτύπου διότι στο παρελθόν είδαμε ότι όταν αναλαμβάνουμε δράση θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή για το συνταξιδοτικό, ενώ μερικές φορές δεν είναι. Τέλος. Ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ηγετικό ρόλο ως προς την εποπτεία του συνταξιοδοτικού για τελευταία χρόνια. Την τελευταία φορά που αναθεωρήσαμε το πλαίσιο ήταν το 2004 για τα συνταξιοδοτικά ταμεία και την ηλικία συνταξιοδότηση. Χρειάζεται περαιτέρω αναθεώρηση. Πασκάλ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ορισμένα στοιχεία από τους πράσινους Συμφωνούμε με πολλές προτάσεις του εισηγητή, ιδιαίτερα ως προς το θέμα αύξησης του δίκτυα απασχολησιμότητας και απασχόλησης μέσα στα πλαίσια του συνταξιοδοτικού. Δεν ξέρω κατά πώς θα πρέπει να το δούμε αυτούσιο αυτό το σύνολο. Υπάρχουν διαφορετικές εθνικές διευθετήσεις, λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές, στο δημοκρατικό. Υπάρχει μια εθνική συλλογιστική δηλαδή ως προς αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει προστιθέμενη αξία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ως προς την ευρωπαϊκή συνεργασία, στο φορολογικό ε, η προστέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξέρω κατά πόσο καθίσταται σαφής, γιατί πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβάλλει τι θα γίνει στα εθνικά συνταξιοδοτικά μέσα στα πλαίσια των ε, γενεολογικών διαφορών. Ε, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα να το δούμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της γενομοδότησης αυτής είναι η αναλογία της δημόσιας άρρωγης και το τι μερίδιο αναλαμβάνει ο δημόσιος τομέας στο συνταξιοδοτικό. Μιλήσαμε και για τον ιδιωτικό τομέα, κάτι το οποίο δεν ευσταθεί, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα κατανομής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ενεργητικού που έχουν συσταθεί, άρα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή τη λογική του ιδιωτικού τομέα, του λογιστικού ιδιωτικού τομέα, στον δημόσιο λογιστικό τομέα. Αλλιώς βάζουμε ένα άλλο στοιχείο, επιπρόσθετο στοιχείο στο δημόσιο χρέος και τα κράτη μπορούν να αλλάξουν τα κριτήρια αυτά που αποτελούν το όλο ζήτημα. Μπορούμε να δούμε το επίπεδο ΑΕΠ, να δούμε την, ε, τα εισοδήματα. Θα δούμε πώς αυτά θα ε, μπορούν να καταστούν μετρήσιμα σε 20-30 χρόνια. Και επειδή αυτό έχει σημασία, στα πλαίσια του δημοσίου χρέους ε, έχουμε μεγάλες αμφιβολίες για το πώς θα μπορέσει να συνεισφέρει στο όλο ε, θέμα. Uh, Είδαμε την άποψη όλων των σκιωδών. Υπάρχουν πολλοί ομιλητές. Uh, uh, και Σκίνερ και Τόμας Μάν. Δεν έχουμε πολύ καιρό. Θα ήθελα να είσαστε ιδιαίτερα σύντομοι. Ο Πίτερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Ζωζ Κούτας για την σχετική εισήγηση και μου έκανε και με θαυμάσιο τρόπο. Έχω τρία σχόλια. Πρώτον, η ΑΙΟΠΑ θα παίξει ένα ρόλο εδώ, Ζωζ, και είναι σωστό να ο νέος οργανισμός ε, συνταξιοδοτήσεων μαζί με τις ιδιωτικές ασφάλειες θα επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορεί ο κ. Καμφά να λέει ότι... Ε, αντίθετα, σε εναρμόνιση. Αυτό θα ήταν απολύτως ακατάλληλο. Για παράδειγμα, στη Γερμανία δίνεται μια ε, απεριόριστη εγγύηση. Το ίδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες, όπου είναι σαφές ότι τα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιμοποιηθούν και οι μηχανισμοί που θα χρησιμοποιηθούν είναι πολύ διαφορετικοί από τον κλάδο των ασφαλίσεων. Και απευθύνω έκκληση να μείνουμε μακριά από αυτό το πραγματικό παγόβουνο του Solvency 2. Ας χρησιμοποιήσουμε τον κλάδο των συντάξεων και τις διατάξεις που υπάρχουν και τους επόπτες, τους οργανισμούς εποπτείας, δηλαδή να δούμε τι χρειάζεται ακριβώς για το συνταξιοδοτικό και όχι για κάτι που μπορεί να τις οδηγεί στην καταστροφή της συντάξης. Επίσης υπάρχουν διαδικασίες και ωφελημάτων και πληρωμών. Δεν χρειάζεται να επιταχύνουμε τα πράγματα αυτά που κάνουμε τώρα. Πρέπει πρώτα να ορίσουμε τις εισφορές και όπως είπε ο Τζόρτζ, θα πρέπει να είναι κάτι ανάμεσα στα δύο. Κάτι που να μπορούν δηλαδή όσες φορές να, πληρώσει, να πληρώσουν οι άνθρωποι. Λοιπόν υπάρχουν τεράστιες συζητήσει πρέπει να γίνουν ακόμα. Όχι όμως μπαίνοντα σε μια ε, πολεμική αντιπαράθεση δηλαδή ε, των συζητήσεων αυτών. Ο Τόμας Μαν ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κούτας. Τόνισε ο κύριος Κούτας ότι σίγουρα έχουμε και προβλήματα αρμοδιοτήτων. Πάντα τα έχουμε αυτά. Τα είδα εγώ και στην Επιτροπή Απασχολήσεως, όπου δεν μας επιτρεπόταν να χρησιμοποιούμε τη λέξη γυναίκες, διότι είναι θέμα της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Τι να πούμε τότε δηλαδή, άνθρωποι μη αρσενικού φύλου. Ε, για μένα <clears throat> είναι αδιαφανή λίγο αυτά. Ότι πρέπει να έχω ομοδιότητα στον τομέα αυτό μου φαίνεται αυτονόητο πέραν των των ακροβατικών αυτοσχεδιασμών. Για, το, για την ουσία τώρα. Έχετε δίκιο κύριε Κούτα στην παράγραφο 4 πρέπει οι χώρες μέλη να έχουν υπόψη στην ευρωπαϊκή διάσταση. Μιλούμε για βιωσιμότητα, μιλούμε για την δυνατότητα μετακινήσεων των εργαζομένων ανάμεσα στις χώρες και να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες να αναλαμβάνουν νέες επαγγελματικές προκλήσεις. Αυτό πρέπει να είναι εξασφαλισμένο. Ταυτόχρονα να περιληφθεί αυτό περισσότερο. Επίσης πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι πλέον, δεν έχουν την παραγωγή τους πλέον σε μία χώρα, αλλά ε, απασχολούν εργαζομένους σε άλλη χώρα. Και μπορεί εν τέλει οι εργαζόμενοι να θέλουν μετά από την συνταξιότησή τους να κατοικήσουν αλλού. Ότι υπάρχει και πρόβλημα χρόνου, ναι, είναι και αυτό σημαντικό. Για το ελάχιστο εισόδημα δεν συμφωνώ της παραγράφου 7. Πρέπει να έχει σχέση με τον κλάδο, με την περιφέρεια, ε, να αξιολογηθεί και να αποφασιστεί από τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Τώρα, οι διαφορές των χωρών μελών, το είπαν και οι προηγούμενοι όλοι, <clears throat> είναι σωστό. Έχουμε διαφορετικές εμπειρίες με αυτό το σύστημα των ε, πολλαπλών πυλώνων και με τις διαφορετικές χρηματοδοτήσεις. Σε πολλούς τομείς έχει αποτυχθεί επιτυχές το σύστημα αυτό, αλλά όχι σε όλους. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να θέσουμε και το ερώτημα. Θα πρέπει να ρυθμιστεί στις χώρες μέλη, αλλά από τους κοινωνικούς εταίρους και νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να παραμείνουμε. Εάν τώρα η οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων που αναφέρεται στην παράγραφο 13 είναι σημαντικό item, αυτό συχνά κρίνεται ασφαλμένα. Δεν είναι περιορισμός του ανταγωνισμού. Ε, εξασφαλίζει την, την ποιότητα της απόδοσης δεν μπορούμε να πούμε όταν υπάρχει η πλέον η ενιαία αγορά δεν θα, μπορεί, δεν θα έχει ε, χώρο η ε, οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων. Για επίσης, όπως είπε και ο Βόλφ προηγουμένως, για την ε, δυνατότητα μεταφοράς των συνταξιωτών δικαιωμάτων. Εάν μειώσουμε όμως εν τέλει το όριο συνταξιοδότησης που τελικά να μην πληρώνεται τίποτα, τότε δεν έχουν νόημα τα ε, συνταξιωτικά συστήματα των επιχειρήσεων. Όπως είπα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να ελέγχουν. Δεν μπορεί το μήνυμα να είναι ότι κάτι που λειτουργεί στις χώρες μέλη δεν μπορεί να λειτουργήσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να είναι απολύτως εξασφαλισμένο τα δικαιώματα των κοινωνικών εταίρων. Υπάρχουν και συντάξεις σε επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται και ε, επιβραβεύουν την πίστη στην επιχείρηση. Δηλαδή επιπρόσθετα λέει η επιχείρηση ε, με τον μισθό σας σας επιβραβεύουμε δίνοντας, προσφέροντας μια εισφορά για το μακροπρόθεσμο συνταξιδοτικό σας σύστημα. Αυτό είναι τμήμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού ε, μοντέλου. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένας τομέας ζωτικός που θα παίξει ρόλο και στις δύο επιτροπές, και της απασχόλησης και την οικονομική. Τώρα για την πρόορη συνταξιοδότηση. Είδαμε ε, στην Γερμανία πώς απορρίφθηκε το σύστημα. Και ότι αναγκάστηκαν να φύγουν εργαζόμενοι από τις επιχειρήσεις με κρατική ενίσχυση, για να δοθούν συντάξει δηλαδή, ταυτόχρονα δεν προσλήφθηκαν όμως νέοι. Θα πρέπει ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στη δουλειά του όσο γίνεται περισσότερο. Πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Και τα πράγματα να μείνουν στα χέρια των χωρών μελών. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Οι βασικέ θεμελιώδει ερωτήσει που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι απαραίτητα σωστέ. Η επικουρικότητα πρέπει να διασφαλιστεί. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μα ήδη λίγο, λέει η προεδρό. και έχουμε και τον Επίτροπο που έρχεται σε λίγο. Δεν μπορούμε λοιπόν να ξεπεράσουμε το όριο των 11. Γι' αυτό να περιοριστείτε σε ολιγόλεπτες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ για Γκαλπέλς. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε νομοθεσία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα θεωρώ ότι είναι επίγον. Έχουμε πολύ διαφορετικά συνταξιοδοτικά συστήματα έχουμε διαφορετικούς ορισμούς και διαφορετικούς κανόνες στα συνταξιοδοτικά μας συστήματα. Εάν συμφωνήσουμε λοιπόν ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινέ, όπως η οικονομική κρίση και οι άλλες, και παγκόσμιες μάλιστα, χρειαζόμαστε ενοποιημένους κανόνες. Σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορες σκέψεις και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί Επειδή τώρα ο προσδόκιμος βίος παρατείνεται, είναι μεγαλύτερος, δεν σημαίνει αυτό ότι γνωρίζουμε αυτομάτως ποιες είναι οι αλλαγές που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες. Η συνάδελφός μου αναφέρθηκε στους τρεις πυλώνες μέσα στο συνταξιοδικό, μέσα στα συνταξιοδικά συστήματα. Είπε επίσης ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη, υπόψη τον κόστος. Γι' αυτό λέω ότι χρειαζόμαστε ενοποιημένη νομοθεσία και ενοποιημένους κανόνες. Υπάρχουν χώρες μέλη που προσφέρουν την επιλογή στους πολίτες τους. Για παράδειγμα, στην Ουγγαρία αυξήθηκε το δημόσιο χρέος σημαντικά, διότι οι πολίτες επέλεξαν ασφαλιστικά συστήματα τα οποία ήταν ιδιαίτερα δαπανηρά για το κράτος. Μάλιστα γι' αυτό το λόγο προσέφηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ουγγαρίας. Η διαδικασία που θα οδηγήσει στην ενοποίηση είναι βέβαια αργή. Γι' αυτό εμεί αποφασίσαμε να περάσουμε σε, από τρεις πυλώνες σε δύο πυλώνες. Ίσως αυτό να μην είναι η σωστή απάντηση, αλλά χρειάζεται να δώσουμε μια επίγουσα απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Έχουμε ένα τεράστιο χρέο και τεράστιο έλλειμμα ταυτόχρονα. Και πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη τη οικονομία. Είναι λοιπόν σοβαρέ οι προκλήσει. Γι' αυτό αποφασίσαμε να λάβουμε επιγόντω μέτρα και να θεσπίσουμε δύο πυλώνες αντί για τρεις. Να παραμείνουν οι πολίτες σε εθελοντικά συνταξιδοτικά συστήματα και να καταργηθούν τα δημόσια. Τι γίνεται όμως με εκείνους οι οποίοι θα φύγουν από τα ιδιωτικά συστήματα και θα περάσουν στα κρατικά συστήματα συνταξιοδότησης. Τι θα γίνουν δηλαδή οι εισφορές τους. Είναι σημαντικό να ζητήσουμε πάντως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση που να οδηγεί σε μια ενοποίηση ή τουλάχιστον ένα βήμα προς μια ενοποίηση και ενοποιημένους κανόνες. Οι τρέχουσες πρακτικές δεν νομίζω ότι θα διευκολύνουν την κινητικότητα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Εσείς έχετε το λόγο. Συγχαρητήρια κύριε Κούτας για την υποβολή της εκθέσεως. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Το ουγγρικό παράδειγμα, το οποίο επισήμανε η συνέδελφός μας, δείχνει ότι η ιδιωτική πλευρά της διασφάλισης των συντάξεων δεν είναι μετέωρη. Έχει γυρίσει την πλάτη του στο μικρόφωνο, δυστυχώς δεν τον ακούμε. Συγγνώμη. Λοιπόν, αναφέρθηκα στην ε, συνάδελφό μου που μίλησε πριν και ήθελα εγώ με τη σειρά μου να πω ότι τα ιδιωτικά συστήματα δεν είναι κάπου στους εθέρες και η απόδειξη είναι πώς έχουν κάνει ράλι και τα χρηματιστήρια ε, ειδικά και στα ζητήματα αυτά. Έχουν συζητηθεί τα ιδιωτικά συνταξιδοτικά συστήματα και παλαιότερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χρειάστηκε να, βγούμε, να αιτιολογήσουμε την ύπαρξη των δημοσίων συντάξεων. Τώρα έχουμε προχωρήσει κάπως από τότε. Για τον Wolf Klintz, για την μεταφορά των δικαιωμάτων. Δεν νομίζω ότι για την αποτυχία της οφείλεται, ε, ευθύνεται το Κοινοβούλιο υπήρξε θέση του Κοινοβουλίου, δεν μπόρεσε όμως να συμφωνηθεί εν τέλει με το Συμβούλιο. Το ζήτημα ήταν να κινηθεί το Συμβούλιο. Ας μην αναζητήσουμε ευθύνες του Κοινοβουλίου. Τώρα, για την ηλικία εισόδου στην σύνταξη. Θα γίνει νομίζω μια ενός είδους ευρωπαϊκή συζήτηση για το θέμα αυτό. Δεν θα μπορούν να είναι μονάχα εθνικά, δεν γίνει μονάχα εθνικά συζήτηση αυτή. Θα ήθελα εδώ να περιληφθεί στη συζήτησή μας ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και στη Γερμανία και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες Πάλι όμως να μην γίνει ιδεολογική συζήτηση στις περισσότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις που γνωρίζω στη χώρα μας δεν υπάρχουν βιομηχανικοί εργάτες πάνω από 50 ετών. Είναι γελίο να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται εφόσον δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια άλλη ε, δόμηση από πλευρά της ίδιας της βιομηχανίας. Χρειάζεται και ε, μια κατάρτιση και μια φροντίδα για την, ηλικία, για την ε, καλή υγεία στην ε, μεγάλη ηλικία που να μην είναι ένα θέμα soft αλλά να είναι θέμα το οποίο να επιβάλλεται και με κυρώσεις. Υπάρχουν και άλλες βέβαια προσεγγίσεις στο θέμα και εκεί προηγούνται οι σκανδιναβικές χώρες. Ο Ρόμπερτ. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι αναρωτιόμαστε ποια είναι η προσθέμενη αξία αυτής της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Ο εισηγητής έχει δίκιο, γιατί νομίζω ότι είναι μηδαμινή, μάλλον δεν ισχύει καθόλου, δεν υφίσταται γιατί μιλάμε για την αρχή επικουρικότητας και αυτό το λέει η ίδια η Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τα συνδιοξιδιωτικά του συστήματα και είναι θέμα προτεραιοτήτων των κρατών μελών. Και είναι θέμα κοινωνικών εταίρων και δεν υπάρχει ενιαίο συνταξιδοτικό οποίο να αρμόζει σε όλους. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής και αυτό είναι το σημείο εκκίνωσης. Όμως στη συνέχεια η Επιτροπή μιλάει για μια ιδιωτικοποίηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Και μιλά για ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Όμως όλες οι ε, αναλύσεις, οι διεθνείς αναλύσεις μιλούν για συστήματα που ε, διέπονται από την κεφαλαιοποίηση. Το Διεθνές ε, Γραφείο Εργασίας λέει ακριβώς ότι μιλάμε για μία αρχή ε, αποταμίευσης και αυτό αυτό που επίσης αναφέρεται είναι ότι ο παράγον της γύρανσης επηρεάζει όλα τα συστήματα κεφαλαιοποίησης. Ο Πιτ Σκίνερ αναφέρθηκε, αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα. Στην αρχή μιλήσαμε για συνταξιοδοτικά ταμεία που ξέραμε τι θα λάβουμε στο τέλος της σύμβασης. Τώρα επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, μιλάμε για συστήματα εισφορών, συγκεκριμένων εισφορών. Ξέρουμε δηλαδή τι καταβάλουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα λάβουμε στο τέλος. και όλοι όσοι υποστήριξαν τα συνταξιοδοτικά ταμεία ως πανάκια είδαν ότι με την επέλευση της κρίσης τα συνταξιοδοτικά ταμεία επλήγησαν γιατί ε, βασιστήκαμε πολλές φορές σε ιδιωτικά συστήματα και τα δύο-τρία τελευταία χρόνια είδαμε μία ε, φθήνουσα πορεία των συνταξιοδοτικών ταμείων. Δηλαδή χάσανε 30% των στοιχείων ενεργητικού, αν όχι και περισσότερο. Αυτό αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Σουηδία που βρίσκονταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Άρα, όποια και να είναι αυτά τα συστήματα, όπως ε, λέει ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μπορντό, τα μία αυτά αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του ΑΕΠ. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο ε, αυτά τα μέσα έχουν συγκεκριμένα ε, απτά αποτελέσματα σε σχέση με το τι έχει κανείς ε, λαμβάνει την επαύριον. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτή την πράσινη βίβλο που είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί όπως είπα και πριν, τα συνταξιοδοτικά συστήματα υπόκεινται στην ε, επικουρικότητα και θα παραμείνουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούτας, δεν έχετε βέβαια τόσο πολύ χρόνο τόσο ώστε να απαντήσετε σε όλα, αλλά πείτε μας δύο λόγια. Ναι κυρία Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Είναι... Όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Όλοι βλέπουν ότι υπάρχουν προβλήματα σε όλες τις χώρες. Προφανώς η αρχή της επικουρικότητας επηρεάζει και τις αποφάσεις μας αλλά αν προ, προσπαθήσω να εξάγω κάποιο συμπέρασμα από τη συζήτηση που έγινε είναι το εξή. αν θέλουμε να κάνουμε κάτι τι πρέπει να δράσουμε δεν πρέπει κάτι να κάνουμε Μέχρι τώρα διαπιστώνουμε προβλήματα αλλά δεν έχουμε λύσεις. Ε, Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν επικοδομητικά και να βρούμε κάποιες λύσεις που είναι βέβαια δύσκολες ε, να βρεθούν αλλά πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουμε. Πρόεδρος, η κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου το μεσημέρι στις 17 Ιανουαρίου στο Στρασβούργο τις, θα τις συζητήσουμε τις τροπολογίες αυτές σε μια έκτακτη συνεδρίαση και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα γίνει ε, στις ε, ε Ιανουαρίου και στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης το Φεβρουάριο αργότερα συγγνώμη, για να μπορέσουν τα πράγματα να πάνε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου ή αργότερα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα και τα λοιπά, η εισηγητής ο κύριος Λάγκεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα για πρώτη φορά συζητούμε τα πολύ σημαντικά αυτά κομμάτια της αγοράς το καλοκαίρι πήραμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες ήταν σημαντικές αλλά σήμερα για πρώτη φορά συζητούμε το θέμα ε, με βάση το κείμενο της Κομισιόν 484 του Σεπτεμβρίου. Αν θέλετε ένα σχόλιο για το κείμενο της Κομισιόν, όντως η Κομισιόν έλαβε υπόψη σοβαρά α, τη θέση του Κοινοβουλίου του Καλοκαιριού. Αυτό είναι πολύ καλό. Η Πρόεδρος θα θυμάται ότι ε, είχαμε μπει και σε λεπτομέρειες. Αλλά η πρώτε Κομισιόν αφήνει εκκρεμή κάποια πράγματα. Και μια και σήμερα γίνει, είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται, θα ήθελα να επαναλάβω κάποιε βασικέ αρχές. Πρώτον, η πρόταση είναι... Ε, συζητήθηκε το Σεπτέμβριο του 2009 στο G20 και εκεί ζητήθηκε διαφάνεια για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα ε, και πάρθηκαν κάποιες σχετικές αποφάσεις. Ή το σχέδιο κανονισμό μου που υποβάλλεται ε, μιλάει για τα παράγωγα, τους κεντρικού αντισυμβαλόμενους και τα αρχεία καταγραφής των συναλλαγών, όμως ε, υπό την... λέει κιόλα ότι πρέπει να γίνει και συντονισμός και συνεννόηση και με τρίτες χώρες γιατί μιλάμε για μια για παγκοσμιοποιημένη οικονομία ουσιαστικά άρα πρέπει να ληφθούν πια μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ε, ξέρετε τι υπογράφηκε, ο, τι έγραψε ο Ομπάμα τον Ιούνιο και εκεί και δόθηκε έτσι μια διετία ε, περιθώρια Βεβαίω οι G20 είπαν ότι στο τέλος του 2012 πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν κανόνες. Άρα ε, οι κανόνες στην αγορά. Άρα μένουν 25 μήνες για να δράσουμε ή να αντιδράσουμε αν θέλετε και μετά αρχίζουν να εφαρμόζονται πολύ συγκεκριμένα, θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται πάρα πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή, αν θέλουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει τον Ιούλιο του 2011 στα τελευταία συνεδρίωση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές του χρόνου να έχει πάρθει απόφαση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως το τι θα κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν το ξέρουμε ακόμη και γι' αυτό δώσαμε εντολή στους δικούς μας εμπειρογνώμονες να ασχοληθούν με, να κάνουν μια σύγκριση μεταξύ του αμερικανικού μοντέλου αν θέλετε ή αυτού που συμβαίνει στις ΗΠΑ και αυτού που συμβαίνει στην Ευρώπη και μέχρι το Γενάρη ζητήσαμε να μας έχουν απαντήσει οι εμπειρογνώμονες τώρα από εκεί και πέρα ε, ο στόχος είναι, γενικότερο στόχος είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι ε, στην αγορά παραγώγων και εκεί ζητούνται μέτρα και τα οποία μέτρα θα μπορούσαν να ήταν παραδείγματο χάρη υποχρεωτικό clearing για κάποια παραγωγότηση ε, τεχνικές προδιαγραφές για την και εποπτεία δημιουργία αρχείων ε, καταγραφής ειδικά κριτήρια για τις, το διμερές clearing συναλλαγών με παράγωγα. Οι, οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται σε μητρώα και ή να δηλώνονται τουλάχιστον σε κάποια κέντρα ε, ε, και οι ρυθμιστικές αρχές ε, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα ε, παρε, ε, να μπουν στα αρχεία αυτά ή στα Μητρώα. Τώρα, έχουμε τα χρηματοπιστατικά ιδρύματα. Εάν η συναλλαγή με παράγωγα δεν γίνει μέσω ενός κέντρου clearing, τότε και γίνει, μέσω ενός κάποιου ιδρύματος τα πράγματα αλλάζουν ε, η Κομισιόν λέει αν δεν πρόκειται για χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τότε υπάρχει υποχρέωση ε, δήλωσης και ενημέρωσης εάν και εφόσον ε, βρισκόμαστε πάνω από ένα κατόφλι. Εδώ, εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχουν ερωτηματικά και κανείς δεν φαίνεται να ε, συμφωνεί ή να μπορεί να εξηγήσει τα δύο κατόφλια που ορίζει εδώ η Κομισιόν ε. και ποια είναι τα κριτήρια τα οποία άμα οδηγούν στον υπολογισμό αυτών των κατοφλίων. Ε, δεν ξέρω Ίσως θα πρέπει να μπει ένα παράρτημα στο κανονισμό που να εξηγεί τα πράγματα αυτά. Αλλά κανείς, κανείς δεν είναι ούτε πρόθυμος να κάνει προτάσεις ούτε να δώσει διευκρινήσεις. Τώρα, λοιπόν, για τα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τις επιχειρήσεις δηλαδή ε, λέει η Κομισιόν ότι υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες υπάρχει δυνατότητα να ασφαλιστούν έναντι των κινδύνων των ρίσκων που υπάρχουν αυτά όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη για, για κάποιους υπολογισμούς αλλά κατά βάση όλες οι συμβα... οι συναλλαγές με παράγωγα πρέπει να μπαίνουν να καταγράφονται σε ένα αρχείο ούτως ώστε να υπάρχει μια συνολική εικόνα της αγοράς άρα πρέπει να οριστούν και διαδικασίες εγγραφής εδώ και υπάρχει και ένα ιδιωτικό ίδρυμα στις Ηνωμένε Πολιτείε που το 2007-2008 μετά την εμφάνιση των προβλημάτων της, το, της κρίσης ας πούμε ε, κατάφερε να κατακτήσει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς ε, που οι Αμερικανοί το εκτιμούν στο 80 περίπου τα 100 και εκεί ε, δηλώνονται τα, τα, οι συναλλαγές. Ρωτούμε λοιπόν, είναι λογικό όλα τα αρχεία για τις συναλλαγές και τα στοιχεία για τις συναλλαγές με παράγωγα να βρίσκονται σε ένα κέντρο αμερικανικό. Θέλουμε να συνεχίσουμε, να ε, αφήσουμε την κατάσταση αυτή να συνεχίσει. Ε, εκτός εάν αν δεν θέλουμε να φτιάξουμε εμείς τα δικά μας τα αρχεία, τουλάχιστον να ζητήσουμε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στη, για τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Στον ιδιωτικό αυτό οργανισμό τον Αμερικανικό. Ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πείσουμε κανέναν να δώσει αυτή την ε, ε, ελεύθερη πρόσβαση, αλλά ε, τι πρέπει να έχουμε και εμείς να κάνουμε με αυτά τα αρχεία. Τώρα για τα κέντρα clearing οι Αμερικανοί έχουν κανόνες και για την διοίκηση αυτών και για τους ίδιους πόρους και τα λοιπά. Υπάρχουν οργανωτικοί κανόνες για πολύ σκληρή διακυβέρνηση και προς αυτά υπάρχουν και στον κανονισμό εδώ που προτείνει η Κομισιόν και λένε, λέγεται επίσης ότι πρέπει να υπάρχει μια ανεξαρτησία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, θα ε, πρέπει να συζητήσουμε εμεί εκτενώς τι γίνεται με τις CCPs. Αυτές οι CCPs υπόκεινται σε κάποια εποπτεία, ζητεί ο κανονισμός τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ίδιο κεφάλαιο, Ά, ίσως πρέπει να αυξηθεί αυτό το ίδιο κεφάλαιο για τα clearing centers. Ένα άλλο θέμα πρέπει να συζητήσουμε είναι η περίφημη interoperability interoperability αυτή η διαλειτουργικότητα ε, αν υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που θέλουν να ε, κάνουν μια τέτοια συμφωνία δια λειτουργικότητας. Βεβαίως με τέτοιου είδους συμβάσεις και συμφωνίες αυξάνονται οι κίνδυνοι στις αγορές παραγόγων. Δεν χρειάζεται να τα πω αυτά. Ε, τώρα ο όγκος της αγοράς αυτής ε, ήταν 650 δις δολάρια στο τέλος του 2008 ε, και γι' αυτό η αγορά αυτή έχει άλλο βάρος για τα μεγάλα κράτη-μέλη και άλλο βάρος για τα μικρα μικρά κράτη-μέλη, όπως τα μικρότερα κράτη-μέλη. Ο, η λοιπόν διαλειτουργικότητας ε, επηρεάζουν διαφορετικά τους μεν και τους δε. Ε, ε, ούτως ή άλλως υπάρχουν εδώ πολλά ερωτηματικά και μεταξύ κρατών μελών το άκουσα και στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου ότι υπάρχουν και για την ομάδα εργασίας του Βουλίου ότι υπάρχουν ε, ερωτηματικά εδώ. Κεντρικό ρόλο παίζουν όπως ε, είπα και πριν τα αρχεία καταγραφής. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Η Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκές αριθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση εκεί ε, πρέπει να υπάρχουν στάνταρ καταγραφής ε, τι γίνεται με την προσθήκη στοιχείων, διαγραφή στοιχείων επίσης, τι γίνεται με την προστασία των στοιχείων, πώς προστατεύονται τα στοιχεία αυτά, είναι ασφαλής η καταγραφή και με ποιο τρόπο προστατεύονται. Έχουμε την υπόθεση SWIFT, τη θυμάστε, ε, εμείς σαν κοινοβούλιο ναι, πρέπει να τη θυμόμαστε πολύ καλά την υπόθεση SWIFT. Ε. Λοιπόν, μην υποτιμούμε την σημασία της προστασίας των στοιχείων εδώ. Η πρόταση του κανονισμού λοιπόν, το σχέδιο κανονισμού, αν μπορώ να το πω εν συντομία, είναι κάτι που το χαιρετίζουμε διότι έχει λάβει που όχι μόνο επειδή έχει λάβει υπόψη αρκετές απόψεις, από τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί, αλλά γιατί για πολύ σημαντικά θέματα ασφάλειας και διαφάνειας είναι βελτιωμένο το σχέδιο αυτοκανονισμού. Μια ιδιαιτερότητα βέβαια του σχεδίου κανονισμού ε, είναι η, ο μεγάλος αριθμός νομοθετικών πράξεων εδώ που εμπλέκονται. Και αυτό το λέει και το Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν την εκτέλεση τόσων νομοθετικών πράξεων να την αναθέτουμε στην Κομισιόν. Το έχουν πει και άλλοι εκτός από μας αυτό βεβαίως. Θα δούμε πώς θα πάνε οι συζητήσεις. Ε, εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε εμείς είναι ότι τελικά βεβαίως το σχέδιο αυτό κανονισμού είναι απλώς ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα πράγματα. Τώρα, χρονοδιάγραμμα προβλέπεται ε, να πάει τέλος Γενάρη, αρχές ε, Φεβρουαρίου ε, το θέμα ξανά εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών γιατί θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας και τις γνώμες των εμπειρογνωμόνων μέχρι τον Ιούλιο θα πρέπει να έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή ούτως ώστε μέχρι το τέλος του 2012 όπως είπα να γίνουν και οι άλλες προετοιμασίες για να μπορέσει να αρχίσει να ισχύει ο κανονισμός. Ε, βεβαίως πολλές εμείς ε, ε, Έχουμε κάνει κάποιες προσωπικές συζητήσεις, έχουν υποβληθεί κάποιες γραπτές προτάσεις, ήρθαμε σε επαφή με τους κοιόδους συζητητές και με τους συνεργάτες τους, όχι μοναχά για να δούμε το χρονοπρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα, αλλά για να δούμε και κάποιες ε, απόψεις και για να ενημερώ, αλληλό, ενημερωθούμε και τελικά φτιάξαμε ένα ερωτηματολόγιο με 10 κύρια ερωτήματα το οποίο το, οποίο το στείλαμε στις, στους, ε, όλους ενδιαφερόμενους ε, με το, την παράκληση μέχρι τις 22 Νοεμβρίου να απαντήσουν. Άρα την περασμένη εβδομάδα πήραμε τις απαντήσεις ε, από μια πρώτη ματιά που είδαμε για τις απαντήσεις είναι σχετικά ικανοποιητικέ. Οι ερωτήσεις αυτές οι 10 αναφέρονται και στα άρθρα και στους ορισμούς και στα κατόφλια που λέγαμε προηγούμενα, άρθρο 7, ε, ζητήσαμε προτάσεις βελτίωσης για την εποπτεία, ιδιαίτερα για τη δημιουργία ενός σώματος βάσει του άρθρου 14 και συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών. Μετά ρωτήσαμε πώς ε, αξιολογείται τη, ε, τον Αμερικανικό νόμο και τη θέση της Κομισιόν ε, σχετικά με τις συμφωνίες και την πρόσβαση στην αγορά των τρίτων χωρών. Τι γίνεται με την διαλειτουργία αυτή την interoperability ε, που σχετίζεται με αυξημένους κινδύνους, τι θα γίνει με τα αρχεία καταγραφής των συναλλαγών, τι πιστεύετε για την, το άρθρο 23, 62, 63 και 67 και τέλος, τι πιστεύετε, κάντε μια γενική ε, κρίση για την πρόταση. Μέχρι χτες το βράδυ είχαμε πάρει απαντήσεις ε, για τα, το ερωτηματολόγιο αυτό πήραμε, 40, είχαμε πάρει 49 απαντήσεις, εκ των οποίων 45 θα μπορούσε να τις ονομάσει κανείς πλήρες γνωμοδοτήσεις τελικά, τις οποίες βεβαίως δεν καταφέραμε να τις αξιολογήσουμε. Ε, ε, περιλαμβάνονται εκεί θέσεις και κρατών μελών και συλλόγων και ενώσεων και άλλων φορέων της αγοράς, ταξιοδοτικά ταμεία κλπ. και κάποιες τράπεζες. Εν μέρη βεβαίως μάλλον βλέπουμε ότι οι γνωμοδοτήσεις αυτές υποβλήθηκαν από συλλόγου συλλόγους ενώσεις και τα και σας παρακαλώ όλους του, τους συναδέλφους ε, να ρίξουν μια ματιά στην αξιολόγηση που θα κάνουμε όταν τέλο πάντων καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό και να βάλουμε στοιχεία στο διαδίκτυο. Τέλος, να κάνω μερικές παρατηρήσεις για το τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Τρεις φορές συνεδρίασε η ομάδα αυτή εργασίας, θα συναντηθεί κι άλλη μια τέταρτη φορά και μετά η Βελγική Προεδρία θα εξάγει κάποια ενδιάμεσα συμπεράσματα. Ε, ε, συστήθηκαν διάφορα θέματα, το κεντρικό clearing και υποχρεώσεις και ε, είπε ότι μπο, μπορεί να υπάρχουν και επιπλέον αποχρεώ... Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούν να επιβληθούν και άλλες υποχρεώσεις ή όχι εάν είναι σωστό να γίνει κάτι τέτοιο από εκεί και πέρα τι γίνεται με τα non-financial derivatives αυτά τα παράγωγα τα non-financial αναφέρθηκα, επικηρύθηκαν τα κατόφλια που ανέφερα προηγούμενα ή συζητήθηκε το θέμα της εποπτείας των CCP και βεβαίως η ε, στο Συμβούλιο υπήρχαν ερωτηματικά, δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε ε, ότι τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου δεν ε, χαίρονται με την καινούργια εποπτική διαδικασία ή αρχή. Από πολλές πλευρές ετέθη το ερώτημα τι θα γίνει άμα δεν μπορούν να συμφωνήσουν, να συμφωνήσει το σώμα αυτό του άρθρου 14 Μήπως ε, έχει πολλά μέλη ε, το σώμα αυτό. Τι γίνεται ε, με τη σύνθεση λοιπόν. Τι γίνεται με τις... χρειάζεται άδεια τραπέζης. Εδώ ο, πολλοί είπαν όχι. Μπήκε το θέμα της κεντρικής τράπεζας. Η CCP ναι, ίσως πρέπει να έχουν λογαριασμό στην κεντρική τράπεζα Τέλος πάντων δεν πάρθηκε απόφαση. Μετά το άλλο θέμα ήταν αυτό των τρίτων χωρών και μπήκε και το θέμα αμοιβαιότητας. Ε, προβλέπεται ένα πλουστευμένο σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης. Ε, είναι ε, ισότιμο αυτό, ισοδύναμο με αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα στην Αμερική, Αμερική είναι πιο δύσκολα από ότι αυτά προτείνει η Κομισιόν μετά μπαίνει και το θέμα των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και φαίνεται ότι εδώ ευθυγραμμιζόμαστε λιγάκι και με την Κομισιόν και με το ο, Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υπομονή σας και περιμένω καινούριε προτάσεις από όλους σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, γιατί οπωσδήποτε ήταν ε, μια πολύ δυνατή παρουσίαση και αυτό που έχει σημασία είναι να εκφραστούν πρώτα οι σκιώδεις. Ο Λεωνάρδο δεν είναι εδώ. Μιλάς εξ ονόματος του Λεωνάρδο. Ευχαριστώ <clears throat> αγαπητές και αγαπητοί φίλοι. Ο σκιώδης συγκητής μας Λεωνάρδο Ντομένιση δεν μπόρεσε να προσέλθει σήμερα λόγω των καιρικών συνθήκων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πρώτα γενικά τον εισηγητή για την περιεκτική και ξεκάθαρη τοποθέτησή του στην αρχή της συζητήσεως εμείς ως σοσιαλιστές και δημοκράτες αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι καταρχήν έχει την υποστήριξή μας για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το θέμα. Βέβαια, κύριε Λάγκεν, αυτό θα ισχύσει μόνο εφόσον ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και δεν θα χάσει το θάρρος του προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτή είναι, αυτός είναι ο βασικός όρος για μας, για τη συνεργασία μας. Χαιρόμαστε που πρόκειται για πρόταση κανονισμού και όχι οδηγίας. Πράγματι όμως, ένα από τα πιο αξιοσημείωτα, αξιοσημείωτα θέματα είναι πόσο μεγάλο είναι το περιθώριο διαμόρφωσης της επιτροπολογίας. Το τονίζω αυτό. Δεν θέλουμε εμείς να παραιτηθούμε από αρμοδιότητες για τις λεπτομέρειες ας πούμε. Ήδη είχαμε τονίσει στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας Λάνγεν ότι δεν μπορούν να βγουν απ' έξω οι αποκεντρωμένοι κίνδυνοι. Θα χρειαστεί να επανέλθουμε και σε αυτούς και στις ασφαλιστικές καλύψεις, καθώς επίσης και αυτά θα συζητήσουμε όταν θα έρθουμε στην οδηγία για την κατάχρηση των αγορών. Τώρα για την ίδια την έγκριση ε, λειτουργίας δεν θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερα περίπλοκη η διαδικασία αυτή. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παίξει έναν ε, ισχυρό ρόλο ο ΕΣΜΑ. Θα κινηθούμε και εμείς προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει ο εισηγητής. Εμείς δεν θέλουμε να αποδυναμωθεί ο ρόλος του ΕΣΜΑ, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα είχε νόημα. Τα ίδια τα CCP πρέπει να έχουν ευρεία πρόσβαση σε ρευστότητα αυτό θα εξαρτηθεί και από, τον, από την διατραπεζική αγορά και από τις παγκόσμιες αγορές. Θα θέλαμε ωστόσο και να συζητήσουμε και με τον εισηγητή και με τους άλλους κοιόδης εισηγητές σε ό,τι αφορά επαρκή κεφαλαιακή πρικοδότηση από την αρχή. Να μην τονίσουμε ιδιαίτερα δηλαδή το προφίλ κινδύνου των CCP και να υπάρξει μια συνολική ρύθμιση. Τώρα, κυρώσεις. Και εδώ θα εξαρτηθεί από την ισχύ του ρόλου του ΕΣΜΑ ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα ίσο, ισότιμο ανταγωνισμό για τα μη χρηματιστηριακά τώρα α, ιδρύματα. Δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε ότι είναι ακίνδυνα. Πρέπει να δούμε και από ποιο είδο δραστηριοτήτων θα προκύψουν κίνδυνοι και από ποιο μέγεθο Σε ό,τι αφορά την, ε, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ Πολιτείες πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ισοτιμία, να μην αποδυναμωθούν οι κανόνες από την πλευρά τους. Θα υποστηρίξουμε τον κύριο Λάγκεν σε αυτό που πρότεινε, το ίδιο ισχύει και για το θέμα της ευρωπαϊκής προσέγγισης για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Θα αρκεστώ για την ώρα σε αυτά. Βλέπετε λοιπόν ότι καταρχήν πορευόμαστε προς μια επικοδομητική συνεργασία με την ελπίδα ότι θα προκύψει ένα στέρεο αποτέλεσμα και μια καλή ρύθμιση. Σημειώνω ότι το ΕΣΜΑ είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγόρων.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 μόνο να σταθώ σε τρία σημεία. Το πρώτο αφορά την πρόσβαση στη ρευστότητα των κεντρικών τραπεζών τη στιγμή που αλλάζουμε τη συλλογιστική μας. Αντί δηλαδή να μιλάμε για διάχυση κινδύνου που οδήγησε στην κρίση, γιατί κανείς δεν ήξερε που βρισκόταν επακριβώς ο κίνδυνος, μιλάμε για μια επανασυγκέντρωση του κινδύνου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι, οι συστημικές αυτές, οι αρχές αυτές αντιμετώπισης του συστημικού κινδύνου δεν θα έχουν πρόσβαση στις, στη ρευστότητα των κεντρικών τραπεζών. Αυτό μας οδηγεί σε πολλά ερωτήματα εναντί του Συμβουλίου και αυτό θα είναι ένα σημαντικό στοιχείο στις συζητήσεις μας. Όπως είπε και ο κύριος Λάγκεν, μας ενδιαφέρει και η διαλειτουργικότητα. Ε, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά από τη στιγμή που μιλάμε για συγκέντρωση των κινδύνων για να μπορέσουμε να τους αποτιμήσουμε καλύτερα, αν μπούμε σε μια ε, λογική διαλειτουργικότητας μεταξύ ρυθμιστικών αρχών, τότε δημιουργούμε ε, μεγαλύτερους κινδύνους, ε, μεγαλύτερους συστημικούς κινδύνους. Διότι δεν ξέρουμε ποιος θα μπορέσει, ποια αριθμιστική αρχή θα μπορέσει να αντιδράσει. Νομίζω λοιπόν ότι η αρχική μας κατευθυντήρια γραμμή είναι να περιορίσουμε τη διαλειτουργικότητα και να θέσουμε δεσμευτικά κριτήρια. Το τρίτο θέμα αφορά το ρόλο των ε, Ευρωπαϊκών Αρχών Κινητών Αξιών και Αγορών, του ΕΣΜΑ, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μία σωστή εποπτεία και προσπαθούμε να ορίσουμε μία ε, αρχή αντιμετώπισης συστημικών κινδύνων γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε μία εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών χωρίς να υπάρχουν αβεβαιότητες μεταξύ ευρωπαϊκού και εθνικού κινδύνου. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να μπορεί να προβεί σε μια συνολική αποτίμηση η ΕΣΜΑ. Σε σχέση τώρα με τις αρχές αυτές, μας ενδιαφέρει να δούμε ποια είναι η θέση και του κεντρικού αντισυμβαλόμενου. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός των διαφόρων κεντρικών αντισυμβαλόμενων δεν πρέπει ε, παρά να προστατεύσει το σύστημα ε, έναντι ενός υπερβολικού κινδύνου και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αναλάβουμε τον κίνδυνο χωρίς όμως να αποτελέσει αντικείμενο ανταγωνισμού. Δηλαδή να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε τους κινδύνους, να τους αποτιμήσει η ΕΣΜΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών μέσα στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής διαιτησίας και αποτίμησης κινδύνου. Αυτές είναι οι γενικές ιδέες που συμμερίζονται αρκετοί συνάδελφοι νομίζω. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε αυτή την αρχή διαλειτουργικότητας μεταξύ ΕΣΜΑ και Συμβουλίου. Thank you, Thank um, Σας ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα σημεία κλειδιά. Νομίζω ότι η καινοτόμος ιδέα του ερωτηματολογίου ήταν εξαιρετική. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι στοιχεία θα φτάσουμε στο τέλος της ημέρας. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ε, ίδιες ιδέες. Γι' αυτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όλοι οι σκιώδεις ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα ήδη από νωρίτερα. Θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την μέχρι τώρα εργασία. Τώρα, ορισμένα βασικά στοιχεία. Είχαμε ένα πολύ εύρωστο ε, έγγραφο από την ε, Κομισιόν και έτσι χρησιμοποιήσαμε και την ε, δική μας έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε τον όρο OTC για όλα τα παράγωγα και δεν μας ενδιαφέρει μόνο το OTC, αλλά όλα τα παράγωγα, διότι οι G20 είπαν ότι θα πρέπει να κινηθούμε ε, μέσα στα πλαίσια μιας μεταρρύθμισης. Θα πρέπει δηλαδή να μιλήσουμε για όλα τα παράγωγα και να μην τα ταξινομήσουμε έτσι ώστε να έχουμε ένα καλύτερο έγγραφο στο τέλος. Ως προς εξαιρέσεις, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλους τους φορείς έτσι ώστε να δούμε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες και να μην αρκεστούμε σε ορισμένα μόνο ε, παράγωγα. Άρα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι οι εμπορικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να ενταχθούν ε, σε έναν κεντρικό μηχανισμό, διότι όταν έχουμε να κάνουμε 160 χρηματιστές, 1600 με συγχωρείτε χρηματιστές, είναι πολύ δύσκολο να τους εντάξουμε κάπου. Άρα θα πρέπει να υπάρχει σωστή ρύθμιση η οποία να ενταχθεί μέσα στους ε, κανονισμούς αυτούς ως προς τους επενδυτές και τις ανησυχίες των επενδυτών που εκφράζονται όχι μόνο στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε όλη την Ευρώπη είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σημείο, μάλλον μία τάση διαχωρισμού στο ανώτερο επίπεδο. Εάν ένας πελάτης θέλει να καταβάλει ένα αντίτυπο αντίτιμο έτσι ώστε να αποχωριστεί, να διαχωρίσει τη θέση του από άλλους πελίτες, δεν βλέπω γιατί να μην μπορεί να γίνει μέσα στα πλαίσια των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Δεν είναι απαγορευτικό το κόστος. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να μπλοκάρουμε αυτή την κίνηση ε, τιμολόγησης, ακόμα και μέσα στα πλαίσια της ρύθμισης. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε μακρύς ορισμούς για τα στοιχεία ενεργητικού που μπορεί να γίνουν αποδεκτά από τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους στα πλαίσια των ταμείων συνταξιοδότησης και των ασφαλιστικών ταμείων γενικότερα. Δηλαδή εκεί υπάρχει ένα ε, περιθώριο με βάση συγκεκριμένες μεταβλητές και θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση για ποια στοιχεία ενεργητικού γίνονται αποδεκτά από τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους διότι αυτή τη στιγμή είναι ε, λίγο συγκεχημένο το μήνυμα και έχει σημασία με ποιους μιλάμε και ποιοι πελάτες αποδέχονται τι. Και αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να γίνει ε, διάκριση σε σχέση με ε, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού. Όταν μιλάμε για συστημικούς κινδύνους θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια προϊόντων, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει ή δεν υπάρχει κίνδυνος, ε, ιδιαίτερα στις αγορές, ε, ε, στις συναλλαγματικές αγορές θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχουν εξοχρηματιστηριακές συναλλαγές. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση συγκεκριμένων προϊόντων, τα οποία βρίσκονται κάταντι της διαδικασίας συμψηφισμού. Δέχομαι τη συνεργασία ΕΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατανοώ ότι ο, διάλογος προωθείται, αλλά επειδή διαχωρίζουμε τα παράγωγα σε τρεις πυλώνες, δηλαδή μύφιτ και κεφαλαιοχικές απαιτήσεις και τα άλλα στοιχεία που δεν συμψηφίζονται δεν θα πρέπει να μας τριμώξουν οι γιατί αυτοί τα αντιμετωπίζουν σαν ένα ενιαίο πακέτο. Εμείς ως προς αυτή τη διάρθρωση δεν θα πρέπει να, να στριμωχτούμε. Δεν χρειαζόμαστε τη λύση των ΙΠΑ μπορούμε να προωθήσουμε δικές μας λύσεις, νομοθετικές λύσεις. Δεν θα πρέπει να μας τριμώξουν οι ΙΠΑ. Κατανοώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ανησυχία, διότι αν είναι κανείς αντισυμβαλόμενος τον ΙΠΑ, δηλαδή αν μιλάμε για την ΕΚΤ ή ε, για ένα ευρωπαϊκό ε, ίδρυμα το οποίο ε, έρχεται σε μια συναλλαγή με το χρηματιστήριο των ΗΠΑ, τότε εντάσσεται στην ομοθεσία των ΗΠΑ ή υπάρχει κάτι αντίστοιχο το οποίο θα περιγράψουμε. Δηλαδή τι μας διέπει ένας ευρωπαϊκός φορέας ή ο αντίστοιχος των ΙΠΑ. Δηλαδή, όταν κανείς έχει συναλλαγές με το χρηματιστήριο των ΙΠΑ, πιο δίκαιο τον διέπει. Και αυτό θα πρέπει να το δουν οι ρυθμιστές και από τη μία πλευρά και από την άλλη, διότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ρύθμιση. Όταν οι ΕΠΑ μας λένε ότι θέλουν να υπάρχει πλήρης ε, ρύθμιση, δεν ξέρω κατά πόσο μιλάμε για κεντρικούς αντισυμβαλόμενους που διέπονται από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ε, ποιο δίκαιο μας διέπει των κεντρικών αντισυμβαλωμένων μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας των ΗΠΑ ή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας γιατί εκτιθέμεθα σε όλα τα παράγωγα και τον είπα και τον είπα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση και έχουμε ενία αντιμετώπιση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ δίκαιοι έτσι ώστε να υπάρχει σωστή ρύθμιση. Ε, um, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι σκιώδης για την ομάδα των φιλελευθέρων και θα ε, παραχωρήσω τη θέση μου γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συμφωνώ με αυτά που προελέχθησαν, δηλαδή ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι πολύ καλή και λαμβάνει υπόψη αρκετά από τα μέτρα τα οποία προβάλλονται και από την έκθεση Λάγκεν αλλά υπάρχουν σημεία που θα πρέπει να διασαφιστούν και τα ανέφεραν και άλλοι ομιλητές Στα θέματα των, του συμψηφισμού και των κεντρικών αντισυμβαλωμένων νομίζω ότι χρειάζεται να δούμε τι μπορεί να συμψηφιστεί για την ε, διαχείριση εξορισμού έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους πελάτες. Και θα πρέπει να δούμε μέσα στα πλαίσια της ρευστότητας των κεντρικών τραπεζών. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε συστήματα όπου οι κεντρικοί αντισυμβαλόμενοι να στέκονται από μόνοι τους. Δεν νομίζω ότι οι φορολογούμενοι μας έδωσαν εντολή, μία εντολή η οποία να μεταφέρει τους κινδύνους άμεσα στους φορολογούμενους μέσω κεντρικών τραπεζών. Και νομίζω ότι διατρέχουμε αυτό τον κίνδυνο, γιατί μιλήσαμε για την διαχείριση κινδύνου. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι να μην λέμε ότι απλώς τα πράγματα ε, γίνονται καλύτερα επειδή ο, τελικός ε, ε, φορέας που δεσμεύεται είναι το κράτος. Το κόστος του συμψηφισμού θα πρέπει να ενταχθεί στον ανταγωνισμό. Εάν η ΕΣΜΑ είναι ε, η, Ευρωπαϊκή αυτή αρχή είναι επικεφαλής αυτής της αρχής, ε, τότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο υφίστανται κίνδυνοι. Ως προς τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους θα πρέπει να έχουμε αποκλειστικές άδειε που να σχετίζονται με την εκτέλεση των πράξεων. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις Ως προς τη διαλειτουργικότητα είναι δύσκολο το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και, όπως σας είπα πριν, δεν θα πρέπει τον κίνδυνο να υπομειστεί ο φορολογούμενος. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ε, για το γεγονός τα παράγωγα είναι ε, μια διεθνής ε, χρηματιστηριακή επιχείρηση. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν οι σωστοί σύνδεσμοι με τα διάφορα ταμεία. Άρα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι στο, για το γεγονός ότι υπάρχουν δύο άκρα σε αυτή την ε, συναλλαγή και θα πρέπει να δούμε σε ποια νομοθεσία υπάγονται οι χ πράξεις. Θα πρέπει να το δούμε μέσα στα πλαίσια των ε, παγκόσμιων στόχων. Αλλά η συλλογή των στοιχείων δεν μας ε, καθιστά ασφαλής. Θα πρέπει να μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε αυτά τα στοιχεία. Άρα η συλλογή στοιχείων θα πρέπει να συνοδεύεται με τις τεχνικές ε, ε, αντιμετώπισης, γενικότερες αντιμετώπισης. Διαφορετικά η συλλογή καθ' αυτή δεν ε, σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ως προς τις ε, ε έχουμε να κάνουμε άμεσα με την υπόθεση Μαρόνι και δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών μπορεί να προβεί σε συστάσεις. Αυτό θα το δούμε. Οι εξαιρέσεις ήδη αναφέρθηκαν για ορισμένους ε, φορείς. Θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό τον κίνδυνο, έτσι ώστε να μην επιβάλλουμε επιπρόσθετες δαπάνες. Δυνάμει του άρθρου 8 αυτό θα πρέπει να μειώσουμε το, τους κινδύνους, να ελαφρύνουμε τους κινδύνους. Γιατί όταν μιλάμε για κεφαλαιουχικές απαιτήσει και για τη σχετική οδηγία θα πρέπει να ενταχθούμε σε αυτό το πλαίσιο. Και να είμαστε σίγουροι τι κάνουμε στο MIFID. Όλα τα άλλα προελέχθησαν Ο κύριος Γκλουτ δεν είναι εδώ. Ο κύριος Τζέντης θα έχει το λόγο ως σκιώδης της Γκου. Ε, ε, ε, Πίτερ Σκίνερ και Βίκη Φόρντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε, πράγματι μιλώ εκ μέρους του κυρίου Κλούτε, ο οποίος είναι ο σκιώδης εισηγητής από την ομάδα μας και ο οποίος δεν κατάφερε να είναι εδώ παρόν. Σε αυτή λοιπόν στην πρώτη ανταλλαγή των σκέψεων που κάνουμε των απόψεων πάνω σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Λάγκεν για την παρουσίαση που έκανε αλλά η βασική μου αρχική μου παρατήρηση είναι ότι η συζήτηση που κάνουμε επί της προτάσεως της Κομισιόν ε, δείχνει ότι η Κομισιόν μάλλον δεν έχει αντιληφθεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα α, ε, σαν ένα μείζον πολιτικό θέμα. Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να παίρνει, με βάση και την πρόταση της Κομισιόν, μόνο μια επιστημονική πλευρά για το είδος και την ποιότητα. Η Κομισιόν ξεχνάει ότι η σημερινή κρίση που βιώνει παγκοσμίω η ανθρωπότητα, η Ευρώπη, αρκετές χώρες, είναι απότοκο της απορρίθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η κρίση χρέους που πρώτα εισέπραξε η Ελλάδα, στη συνέχεια η Ιρλανδία, σε λίγο δεν ξέρω ποιες άλλες χώρες, είναι αποτέλεσμα της δράσης των μαφιόζων της αγοράς. Και η Επιτροπή με την πρότασή της δείχνει να μην το καταλαβαίνει, να μην θέλει να το αντιμετωπίσει και θεωρεί ότι με μέτρα εποπτείας, χαλαρής όμως εποπτείας, δεν θα ξαναγίνει το 2008. Εν πάση περιπτώσει, αλλιώς θα έπρεπε να κινηθεί η Επιτροπή, αλλιώς θα έπρεπε να τεθεί το θέμα, όμως αυτό έχουμε, με αυτό συζητάμε. Συμφωνώ λοιπόν ότι είναι αναγκαία η εγκατάσταση, αναγκαία η εγκατάσταση κεντρικά αντισυμβαλωμένων ε, φορέων. Όμως, επειδή πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στα μέτρα υποπτίας, θα πρέπει να πούμε ότι αν αυτοί οι κεντρικά αντισυμβαλλομένοι φορείς αποκτήσουν τέτοιο ρόλο, όπως τηρημένων των αναλογιών ή οίκοι αξιολόγησης και δημιουργήσουν καινούργια κρίση, θα πρέπει αυτό δεν μπορούμε να το μαντέψουμε αλλά προφανώς χρειάζεται ισχυρή εποπτεία και με αυτή την έννοια συμφωνούμε σε μέτρα αυτή τη κατεύθυνση. Δύο παρατηρήσει επί τη ουσία για να μην σα κουράσω στην πρώτη. Το πρώτο, ότι αυτό το πεδίο εφαρμογή τη εποπτείας, νομίζω υπόθηκε και από άλλου συναδέλφου και τη συναδέλφισσα, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα μη τυποποιημένα προϊόντα, αυτέ τι διάφορε καινοτομίε που βρίσκει ο χρηματοπιστωτικός τομέας, εφευρετικότατο κατά τα άλλα, για να ξεφεύγει από του κανόνε. Και αυτό παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα, έχει σχέση και με την αρχική μου παρατήρηση και νομίζω ότι όλοι εδώ συμφωνούμε. Και η δεύτερη, ότι μια ισχυρή εποπτεία, για την οποία δουλεύουμε ε, και η σκέψη αυτή, ξαναλέω, ακούστηκε και από άλλους συναδέλφους, θα πρέπει να ελέγχει και την εκαθάριση του κεντρικού αντισυμβαλόμενου που βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Ένα καθεστώς εξαιρέσεων θα δημιουργήσει ανισορροπίες και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση οι δικέ μας προτάσει θα πρέπει να προβλέπουν οι δραστηριότητες αυτές να ρυθμίζονται και να εποπτεύονται από, κεντρικές, από ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Θα ήθελα να περιουστώ σε αυτές τις πρώτες παρατηρήσεις και θα συμβάλλουμε στην προσπάθεια που κάνει ο συνάδελφος και ο κύριος Κλούτε ως ε, σκιώδης συζητητής να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Uh, thank Σας ευχαριστώ. Εσείς τώρα κύριε Σκίνερ. Εγώ ευχαριστώ τον Βέρνερ Λάγκεν για το έργο του. Άκουσα και άλλους που συμφωνούν ότι είναι εντελεχέστατη αντιμετώπιση του θέματος. Τώρα, για την έγκριση για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, τα CCP. που από το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει εφόσον πρόκειται για μια κοινή, κοινή ε, γνωμοδότηση θα χρειαστεί ομοφωνία. Αν δεν καταφέρουμε τέλο πάντων να υπάρξει ομοφωνία και ξέρουμε οι νομοθέτες πώς δρούν, είναι πολύ δύσκολο και οι 27 να συμφωνήσουν. <clears throat> θα πρέπει να παρεμβαίνει ο ΕΣΜΑ με απλή πλειοψηφία εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Ορισμένοι θα συμμετέχουν θα είναι οι κεντρικοί τραπεζίτες. Αν λοιπόν κάποιος πει όχι, πού πάμε από εκεί και πέρα. Υπάρχουν λοιπόν περιπλοκότητες στο σύστημα που θα καταστήσουν πολύ δύσκολη την έγκριση μιας κοινή γνωμοδότησης. Έχοντας περάσει και τόσους μήνες για την εκπόνηση των διαδικασιών αυτών που πρόσφατα υπερψήφισε το Κοινοβούλιο για να προχωρήσει η συζήτηση στα σώματα με διαδικασία διαφοράς. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πρώτα αυτό πριν πάμε να επινοήσουμε κάτι καινούριο. Τα λέω λοιπόν αυστηρά στην ε, Κομισιόν. Πήγανε να περάσουν κάτι, αλλά το είδαμε, το πρόσεξα θα πρέπει να προσέξουμε πολύ να μην περάσουν πράγματα από την πίσω πόρτα από αυτά που αρέσουν στην Κομισιόν και που είναι αντίθετα με αυτά τα οποία πρόσφατα ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε και τις, μακρο, τα, τις αποταμιεύσεις. Η Κέι σωστά είπε ότι το πρόβλημα και ιδίω για τις συντάξεις μιλάμε δηλαδή για χαμηλού κινδύνου και υψηλής ρευστότητα αποθεματικά. Είναι σημαντικό να ακούσουμε γιατί ο κόσμος συχνά μιλάει υποκριτικά κάπως λέει ότι πρέπει να είμαστε φιλοευρωπαίοι και για άλλα θέματα δεν δέχονται τους ίδιους κανόνες. Ζητούν εξαιρέσεις επί εξαιρέσεων. Ας είμαστε λοιπόν λογικοί στο πώς θα το προσεγγίσουμε το θέμα. Χρειάζεται ένα συμβασμός, Βέρνερ Λάγγεν και να δω πώς θα τον επιδιώξεις. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Λάγγεν για την πολλή δουλειά που έκανε δύο σύντομα τεχνικά θέματα. Η σχέση δηλαδή για την, ε, με την οδηγία κεφαλουχικών απαιτήσεων. Τι είναι πρώτα liquid asset, ε, ρευστό ε, περιουσιακό στοιχείο και όπου θα είναι αυτό δηλαδή όπως και θα γίνεται η συναλλαγή. Τώρα, στην οδηγία για τις κεφαλουχικές απαιτήσει. είχαμε μια μεγάλη συζήτηση, μάλιστα σε αυτή την αίθουσα εδώ, σχετικά με το τι είδους ε, στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να διαθέτει η τράπεζα. Γιατί για να αντιμετωπιστούν απαιτήσει της ε, νέας ε, συμφωνίας της Βασιλείας δεν υπάρχει επαρκή ρευστότητα σε όλο τον κόσμο για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσει της Βασιλείας 3. Για το λόγο αυτό κάνουμε τη συζήτηση σχετικά με καλυμμένες ομολογίες ή ε, διασφαλισμένες, καλυμμένα ομόλογα μάλλον και ούτω καθεξής. Από πού θα βρεθεί αυτή η ρευστότητα λοιπόν στην Βασιλεία 3 έχουν μια περίοδο 8 ετών οι τράπεζες για να εμφανίσουν αυτά τα νέα καλάθια ρευστότητας. Από πού θα βρεθεί όμως αυτή η ρευστότητα από τις αγορές. Αυτό που χρειάζεται είναι να κινηθεί η συζήτηση στο ίδιο επίπεδο και να σκεφτούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτής της σημαντικής αλλαγής στην ευρύτερη οικονομία. Το άλλο θέμα είναι για τους τελικούς χρήστες και πώς θα αντιμετωπιστεί στη συζήτηση για τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει. Θα είναι κρίμα αν έχουμε αποφασίσει όταν, για να υπάρχει η κάλυψη αυτή, πώς ε, θα την εγκρίνουμε και θα υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ Πολιτείες γιατί εκεί είναι πολύ πιο ρευστή αγορά στα παράγωγα. Εκεί ο αντισυμβαλόμενος μπορεί να κάνει hedging ενός τμήματος πολλώντας ένα παράγωγο πίστης. Εδώ δεν έχουμε τέτοια αγορά παραγωγών στην Ευρώπη και επομένως ίσω να μην μπορεί να γίνει η αντίστοιχη κίνηση. Είναι περίπλοκο και τεχνικό το θέμα, το κατανοώ αυτό, αλλά ίσως η διαφορά που θα προκύψει να είναι πάρα πολύ σημαντική. Η ομάδα εργασία της Κομισιόν που επεξεργάζει το θέμα καλά θα ήταν να συνεργαστεί με αυτούς που εργάζονται επί του CRD4 και να δουν εάν μπορεί να, υπάρχει, να υπάρχουν διαφορετικές διατυπώσεις για τα ευρωπαϊκά ε, ιδρύματα που κάνουν την ίδια δουλειά όπως ε, στις ΗΠΑ. Η Κομισιόν είναι παρούσα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σύντομα. Ζαν Πολ, ο τελευταίος ομιλητής. Θα ήθελα ως τελευταίος ομιλητής πριν από τον Επίτροπο να ευχαριστήσω τον κύριο Λάγκεν γιατί αυτό δεν το κάνω από συνήθεια, το εννοώ γιατί μέσα από τη διαδικασία διαβουλεύσεων έφτασε σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα ως προς το πεδίο εφαρμογής. Δεν θα πρέπει να χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο ε, έχει σχέση με την εμβέλεια της ε, οδηγίας. Δεν θέλουμε να ακούμε τα άσχετα μυρολόγια. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε την αγορά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω ότι η πρόταση της ε, Επιτροπής ε, είναι θετική και εξισορροπημένη και μίλαμε για απτές προτάσεις στην έκθεση πρωτοβουλίας. Δέχομαι αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής ε, ο, και θα πρέπει να δούμε τι μπορεί, πώς μπορεί να συνεισφέρει η ΕΣΜΑ διότι από τον Μαρόνι έχει παρέλθει πολύς χρόνος και ως προς τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ε, βρέθη μία λύση. Άρα η ΕΣΜΑ θα πρέπει να έχει τις σωστές αρμοδιότητες, κατάλληλες αρμοδιότητες. Θα πρέπει να υπάρχει και αμοιβαιότητα, ο Βέρνερ Λάγκεν το τόνισε, δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς, θα πρέπει και είπα να μην ε, προβάλλουν αυτόν τον ευφύ προστατευτισμό και ε, να μην μπορούμε να μπούμε στην αμερικανική ε, αγορά. Νομίζω ότι αρκέστηκα στο 1,5 λεπτό και σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο και πάλι στον εισηγητή για να απαντήσει. Κύριε Πρόεδρε, προτιμούσα μάλλον να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ σημείωσα όλες τις παρεμβάσεις των συναδέλφων μου, θα τις αξιολογήσω. Θα προτιμούσα να έλεγε κάτι ο κ. Πίρσον. Patrick, θέλετε να λάβετε το λόγο. Πολύ σύντομα, ωστόσο. A few points, Madam Λίγα θέματα, κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση της Κομισιόν έχει εμπνευστεί σε μέγα βαθμό από την έκθεση και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου καθώς και από την εργασία του κ. Λάγκεν και των άλλων συναδέλφων του. Ευχαρίστως προωθούμε το, την εργασία αυτή περαιτέρω, εξαιρετική δημόσια διαβούλευση και εμείς θα προπαρασκευάσουμε και τις ε, απαντήσεις ε, της ε, δημόσιας διαβούλευσης που θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα μας. Άρα μέχρι τώρα καλή συνεργασία. Τώρα, για το πεδίο εφαρμογή, ορισμένα ενδιαφέροντα θέματα που ακούστηκαν για τα παλαιά παρόαγωγα, όχι μόνο τα λεγόμενα OTC, τις εξοχρηματιστηριακές συναλλαγές. Τώρα, για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, μας άρεσε που με την εξαίρεση των collateral των ενεχείρων θα, θα συμφωνήσουμε δεν θα αδειάσει η ρευστότητα από την οικονομία με τον τρόπο αυτό. Τρίτο θέμα, ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στις εξελίξεις της ΗΠΑ. Η πρόταση της Κομισιόν εγκρίθηκε ταυτόχρονα με το Dot Frank. Τώρα αρχίζουν να φαίνονται λεπτομέρειες από τις Αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές. Πρέπει να δούμε και εμείς να είμαστε τουλάχιστον ισοδύναμοι σε προδιαγραφές και σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες των ρυθμιστών μας. Μας ενδιαφέρει η συγκριτική εργασία λοιπόν που κάνει η Επιτροπή σας. Για την διαλειτουργικότητα συμφωνούμε ότι υπάρχουν έξτρα κίνδυνοι, συμφωνούμε απολύτως, γι' αυτό η πρόταση της Κομισιόν είναι περιορισμένη, δεν καλύπτει τα παράγωγα, δεν θα πρέπει να καλύπτει και τα παράγωγα. Ε, ε, καλύπτει μόνο τα λεγόμενα cash equities και μόνο εφόσον συμφωνήσουν όλοι οι ρυθμιστές. Νομίζω λοιπόν εδώ πατάμε γερά στο έδαφος. Τώρα, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών. Ακούσαμε τις απόψεις πολλών συναδέλφων σας ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα διεθνές, παγκόσμιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή ε, προσέγγιση. Ακούσαμε τον κύριο Σκίνερ ότι υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν. Συμφωνούμε απολύτως ότι δεν θέλουμε κοινή γνωμοδότηση της ΕΣΜΑ και ούτε περιλαμβάνει τέτοια στο άρθρο 13 η πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω ότι συμφωνούμε εδώ με τον κύριο Σκίνερ. Ένα τελευταίο σχόλιο. Το σύστημα δηλαδή που ε, θεσπίζουν τώρα τα θεσμικά όργανα. Εμείς απαιτούμε όλες οι επιχειρήσεις να περάσουν από αυτούς τους κεντρικούς συμβαλόμενους. Πολλοί βουλευτές είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην ρευστότητα των κεντρικών τραπεζών. Ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Να έχουμε δηλαδή καλύτερη επισκόπηση του συστημικού κινδύνου που θα προκύψει. Να έχουμε ξεκάθαρη επισκόπηση των CCP και των τρόπων με τον οποίο ε, ε, συνεργάζονται και να γίνουν και stress test για τους ε, κεντρικούς συμβαλόμενους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είμαι βεβαία ότι κατανοήσατε και τις απόψεις που εκφράστηκαν εδώ σχετικά με την οδηγία για τις κεφαλαιοχικές απαιτήσει και ίσως βοηθήσετε ώστε να περάσουν και στην Κομισιόν. Κύριε Λάγκαν, είστε ευχαριστημένος από τις απαντήσεις αυτές. Εντάξει, ευχαριστώ. Όπως είπε ο εισηγητής, το σχέδιο εκθέσεως θα είναι διαθέσιμο περί τα τέλη Ιανουαρίου, όταν θα λάβει δηλαδή την έκθεση των εμπειρογνωμόνων για τα θέματα που έχει θέσει και αναμένουμε προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών να είναι στις 15 Δευτέρου, εξέταση των τροπολογιών στις 15 Μαρτίου, ψηφοφορία στις 23 Μαρτίου. Αυτό είναι το προσωρινό χρονοδιάγραμμα. Όπως είπε ο εισηγητής, πρέπει να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια το αργότερο, τον Ιούλιο, 7ο μήνα. Τώρα θα προχωρήσουμε στο θέμα υπαριθμών 5 και με μεγάλη, με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον ε, Επίτροπο κ. Σέμετα, Επίτροπο για την Φορολογία και την Τελωνιακή Ένωση, Λογιστικό Έλεγχο για Καταπολέμηση της Απάτης για τον διαθρωμένο διάλογο για τις πολιτικές προτεραιότητες που ε, κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι αρμόδια για, μια, για ένα ε, τομέα όπου εμείς έχουμε αρμοδιότητα. Θα δώσω ε, αμέσως τον λόγο στον Επίτροπο. Όσοι παρακαλώ επιθυμείτε να εξέλθετε, μπορείτε να συζητήσετε έξω από την αίθουσα. Σας παρακαλώ. Μπορείτε να αποχωρήσετε ήσυχα. Κύριε Επίτροπε. Κυρία Πρόεδρε, Θυμάμαι την, ε, τη συζήτηση που κάναμε τον Ιούνιο όταν ε, ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίως και με τις συζητήσεις που έγιναν έκτοτε ε, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει ε, τρομακτική διαφωνία μεταξύ ε, ημών και ημών. Να σας πω όμως τι έγινε και να τι ε, πρωτοβουλίες θα αναλάβουμε του χρόνου. Το οικονομικό ε, περιβάλλον αυτή τη στιγμή ε, είναι τέτοιο ούτω ώστε να είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητηθούν ε, θέματα κοινή φορολογικής πολιτικής παραδείγματος χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είπαμε όμως πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και όπως είπαμε και στην ε, ομάδα για την φορολογική πολιτική και όπως λάβαμε και την περασμένη εβδομάδα ε, πρέπει να γίνουν οι συζητήσεις αυτές και μελλοντικά θα πρέπει να ασχοληθούμε με καταναλωτικούς φόρους, φόρους για την προστασία του περιβάλλοντος, εταιρικούς φόρους και να συζητήσουμε και θέματα καταπολέμησης, φοροδιαφυγής και απάτης. Σήμερα θα σας αναφέρω ποια είναι οι νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες για του χρόνου. Μαζί με τον κύριο Μπαρνιέ ε, έγιναν κάποιες προτάσεις και υιοθετήθηκαν κάποιες από αυτές μες στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Καλή φορολογική πολιτική και εναρμονισμένη παρόμοια αν θέλετε στην Ευ... σε όλα τα μέρη της Ευρώπης φορολογική πολιτική ε, θα είναι κάτι που θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες το αυτή τη στιγμή βεβαίως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να άρουμε τα εμπόδια αυτά και να κάνουμε πιο εύκολο τη διασυνοριακή συνεργασία των επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να λειτουργήσει καλύτερα η κοινή αγορά. Μέχρι την Άνοιξη ελπίζουμε να κάνουμε πρόταση για τον εταιρικό φόρο. Ε, επίσης πιστεύουμε ότι θα ε, μπορούσαμε να ε, στον τομέα των εταιρικών φόρων να ε, κάνουμε και επιμέρους προτάσεις πιο πρακτικές που να μπορούσαν να εφαρμοστούν από τα διάφορα κράτη μέλη. Δεύτερο θέμα, ΦΠΑ. Εδώ υπάρχουν προκλήσεις τις οποίες πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Βεβαίως ο κύριος Κάσα δεν ξέρω α, υπέβαλε, ήταν ο εισηγητή για μια έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό που εγκρίθηκε την περασμένη ολομέλεια, την περασμένη εβδομάδα. Ε, ξέρουμε ότι δεν συλλέγεται γύρω στο 12% του ΦΠΑ που οφείλεται. Αυτό ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως επιχειρήσει τα στα διάφορα κράτη-μέλη. Τρίτο θέμα. Η Κομισιόν paper on innovative financing in April. Ε, τον, για την φορολόγηση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Τα θέματα αυτά τα συζήτησε η Κομισιόν στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι η κυρία Ποδηματά για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας ε, ετοιμάζει μια έκθεση. Παρακολουθούμε μεγάλο ενδιαφέρον τη δουλειά αυτή ε, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα επιμένουμε στην προστασία του πολίτη στην προστασία από τη διπλή φορολογία ε, και ξέρουμε ότι πραγματικά με τις παρακρατήσεις φόρων ε, και τα λοιπά ιδιαίτερα υπό ότι μέσα στην μια περίοδο κρίσης όπως το ο πολιτής υποφέρει για τα δικαιώματα, για τα, τους τόκους και τα λοιπά. Αυτά είναι επίσης θέματα που αφορούν άμεσα το πολίτη και τα οποία θα συζητήσουμε το χρόνο Την περασμένη εβδομάδα ε, τον περασμένο Ιούνιο ελέγχθη επίσης ότι το σύστημα που ισχύει αυτή τη στιγμή δεν στηρίζει, δεν, δεν μας δίνει χένια για το ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι βεβαίως υπό συνθήκες κρίσης δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά του χρόνου προθυτίθεμε να υποβάλω ε, μια πρόταση στους, υπόλ, στους συναδέλφους μου μου ε, επιτρόπους. Πέρσι εγκρίθηκε ένας κανονισμός του Συμβουλίου που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή όσον αφορά του ΦΠΑ συγκεκριμένα. Όμως Ελπίζουμε λοιπόν του χρόνου να εφαρμοστούν οι διατάξεις του κανονισμού αυτού και το Eurofisc και η αυτόματη πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία να λειτουργήσουν επίσης. Ε, η Βελγική Προεδρία έκανε πολύ καλή δουλειά και πιάρθηκαν πρόσφατα αποφάσεις στο Συμβούλιο που εξασφαλίζουν πρόοδο. Well, I would wish but are nevertheless progressing. Επίσης, α, ένα άλλο θέμα είναι το εξής. Ε, κανείς δεν πιστεύει ότι ε, για ε, τα επιμέρους μέρη του πακέτου που απάπτονται των φορολογικών θεμάτων ε, μπορούν να συζητηθούν χώρια. Ε, για την οδηγία υπάρχει μεγάλη υποστήριξη. Το Δεκέμβρη θα συζητηθούν λοιπόν όλα τα θέματα μαζί. Ε, στην επόμενη προεδρία την, της Ουγγαρίας θα πρέπει ε, να συζητηθούν επίσης συμφωνίες για την καταπολέμηση της με τρίτες χώρες. Είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την, ε, τον αθέμητο ανταγωνισμό. Υπάρχει το θέμα επίσης του λίχτενστάν και τέτοιου είδους φορολογικών παραδείσων. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτές τις χώρες. Υπάρχει και το θέμα του κώδικα δεοντολογίας που θα συζητηθούν στην επόμενη συνάντηση της ομάδας για την οικονομική πολιτική και κλείνοντας να πω μερικά πράγματα για την πολιτική εξόδου από την κρίση. Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή καλούνται να εφαρμόσουν συστήματα δημοσιονομικού περιορισμού για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Ο, είμαι πεπισμένος όμως ότι ότι 27 διαφορετικές προσεγγίσεις δεν θα δώσουν καλά αποτελέσματα. Πιστεύουμε στην ομάδα φορολογικής πολιτικής ότι θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση για να πιστούν τα κράτη-μέλη για να δούμε τι μπορεί να γίνει κοινά από τα κράτη-μέλη στο μέτρο της φορολογικής πολιτικής. Βεβαίως α, χαιρετίζουμε τα αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στα διάφορα κράτη-μέλη για την έξοδο από την κρίση. Θα τα μελετήσουμε περαιτέρω και θα δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε μια ομοιόμορφη κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. And of Σας ε, αποστέλω μία επιστολή για να λάβετε μέρος στην στην ε, καινοτόμο χρηματοδότηση που θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου. Να προσέλθετε δηλαδή στην ακρόαση αυτή της 10 Ιανουαρίου για την καινοτόμο χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση καινοτομία σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, ερωτήσεις τώρα. Θα έχουμε μία ερώτηση, μία απάντηση. Να είσαστε σύντομοι. Δεν θα δεχτώ πολλαπλές ερωτήσεις από έναν διότι δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ να είσαστε λογικοί έτσι ώστε ο Επίτροπος να μπορεί να απαντήσει. Uh, uh, uh, Jose Garcia Magallo, Annie Podimata, Udo Bullman, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzes, Provence Beres, Sven Giegold, Philip Lamberts, Wolf Klintz and Sophie Intveld. If there's anybody else... Αυτός ήταν ο κατάλογος. Αν, είναι, αν υπάρχει και κάποιος άλλος να μου το πει τώρα. Όχι, εντάξει. Το λόγο έχει. Well, thank you, Commissioner. I'll be very specific on, my question to save time. Η Αιλίν, θα ήθελα να σας μιλήσω για την τρίτη προτεραιότητα, για την φορολόγηση των, του χρηματοπιστωτικού τομέα. Γιατί δεν είδατε καν τι γίνεται με τον Ευρωπαϊκό Φόρο Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πρόσφατη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ, όπου βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν στην Ευρωζώνη, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε 20 δις ευρώ. Δεν πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να αποποιηθείτε αυτό τον φόρο χωρίς να δείτε πώς έχουν οι μελέτες γιατί ε, αρνηθήκατε αυτή την επιλογή τη στιγμή που δεν έγινε μια μελέτη αντικτύπου εφόσον το Κοινοβούλιο ζήτησε κάτι τέτοιο. Δηλαδή να δείτε τι γίνεται με τον Ευρωπαϊκό Φόρο Χρηματοπιστών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Να το σκεφτείτε δηλαδή και να δείτε ποια είναι αυτή η επιλογή, πώς έχει αυτή η επιλογή, ακόμα κι αν είμαστε αρκετά περιορισμένοι. Δεν πρέπει να το απορρίψετε όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Θα ήθελα να πω ότι πριν την ανακοίνωση προβήκαμε σε μία λεπτομεριακή ανάλυση για την χρηματοδότηση της καινοτομίας και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς έχει αυτή η ανάλυση, πώς προβαίνουμε σε αυτή την ανάλυση. Και σε αυτό το στάδιο δεν βρήκαμε κανέναν τρόπο που θα μας επιτρέψει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή η φορολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα ε, είναι επιζήμια στον ανταγωνισμό. Γι' αυτό η ίδια η ανακοίνωση τονίζει ότι θα συνεχίσουμε να προωθούμε τον φόρο ε, συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ δεσμευτήκαμε ως Επίτροπη και παράλληλα θα ασχοληθούμε και με τον, την φορολόγηση της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας. Επίσης, θα δούμε πώς θα προωθήσουμε την φορολόγηση του των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών με βάση μελέτες αντικτύπου. Άρα μιλάμε για μια γενικότερη, γενικότερη αποτίμηση και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ε, μια μελέτη αντικτύπου που θα ορίσει την περαιτέρω φορολόγηση. Ο Ιωσέφ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Στα πλαίσια του σχεδίου διάσωσης της ε, Ιρλανδίας συζητήσαμε για τον φορολόγηση αυτή χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Νομίζω ότι θα μας μιλήσετε για την ενιαία φορολογική βάση για τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μέσα στα πλαίσια του ε, κώδικα καλής συμπεριφοράς Θεωρείτε ότι το 12,5% αποτελεί στρέβλωση στον ανταγωνισμό. Well, I think, uh, first... Απάντηση. Θα πρέπει να τονίσω ότι ο παρόν κώδικας συμπεριφοράς έχει σαφή κριτήρια Υπάρχουν πέντε κριτήρια τα οποία ορίζουν τις πρακτικές που θεωρούμε βέλτιστες φορολογικές πρακτικές, καθώς και τους δείκτες φορολόγησης. Οι δείκτες φορολόγησης δεν εμπίπτουν στα κριτήρια φορολογικού ανταγωνισμού. Είπα στην αρχή ότι θα δούμε το παρόν σύστημα φορολόγησης των επιχειρήσεων με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς και αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο στην ομάδα φορολόγησης, αποτίμησης φορολόγησης. Είδαμε πολλές εξελίξεις πρόσφατα ως προς την ε, φορολόγηση επιχειρήσεων. Και θα το δούμε και περαιτέρω τη στιγμή που δεν συμπίπτουν απόλυτα τα φορολογικά συστήματα. Και θα δούμε και τα άλλα ανακύπτοντα ζητήματα που είναι απότοκα αυτού του φαινομένου. Θα μπούμε λοιπόν σε ενδελεχή συζητήσεις ως προς τον κώδικα συμπεριφοράς, καθώς και τα κριτήρια που πρέπει να τον διέπουν. Και θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό περαιτέρω στην επόμενη ομάδα αποτίμησης φορολόγησης τώρα. Ως προς τους ε, φορολογικούς δείκτες γενικότερα, Είπα εξ αρχής και έχω πει πολλές φορές ότι δεν νομίζω ότι οφείλουμε να εναρμονίσουμε τον εταιρικό φόρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τον φόρο επιχειρήσεων, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες δομές ανταγωνισμού μέσα στο εταιρικό σύστημα που είναι ε, υγιείς, που αποτελούν υγιείς μηχανισμούς. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιλύσουμε όλα μας τα προβλήματα μέσω δικτών, αυξάνοντας δηλαδή τους δίκτες φορολόγησης, τους συντελεστές φορολόγησης. Εγώ προωθώ την εναρμόνιση του εταιρικού φόρου, αλλά σας είπα στην εισήγησή μου ότι θέλουμε να εναρμονίσουμε το CCTB και θα έχουμε μία ενδελεχή συζήτηση επί του θέματος εδώ στο Κοινοβούλιο. Σε σχέση με τους συντελεστές φορολόγησης πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποτιμήσουν τα φορολογικά του συστήματα, λαμβάνοντας υπόψη και το μακροοικονομικό περιβάλλον για να αποφασίσουν ποιος είναι ο σωστός φόρος υπό τις ε, μακροοικονομικές συνθήκες. Ευχαριστώ. Ιάννη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας κύριε Επίτροπε. Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Θα συνεχίσω ε, στην κατεύθυνση του ερωτήματος που υπέβαλε η συνάδελφος η Αλίνη Μακάρθη. Στην ανακοίνωση που ε, παρουσιάσατε τον περασμένο Σεπτέμβριο για την ε, φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού παρουσιάζει δύο βασικές εναλλακτικές προτάσεις για τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τη θέσπιση φόρου επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, καταλήγει ουσιαστικά στο συμπέρασμα ότι ο πρώτος είναι κατάλληλος για να εφαρμοστεί στο παγκόσμιο επίπεδο και ο δεύτερος στο ευρωπαϊκό. Ε, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ρωτήσω πώς χωρίς να έχει προηγηθεί μια ενδελεχής μελέτη σκοπιμότητας καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το συμπέρασμα. Ε, δεν μοιάζει λίγο σαν να έχει προαποφασίσει η Επιτροπή προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί χωρίς να έχει, γίνει, ε, να έχει προηγηθεί μια ενδελεχής μελέτη επιπτώσεων. Και το δεύτερο, αφού η ίδια η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της αναγνωρίζει ότι στην περίπτωση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, υπάρχει ένας ισχυρός ρυθμιστικός ρόλος και επίσης τα έσοδα είναι πολύ περισσότερο συγκεντρωμένα από ότι στο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Παρόλα αυτά, ε, καταλήγει στο συμπέρασμα ε, ότι προκρίνει για το ευρωπαϊκό επίπεδο τον φόρο επί των ε, χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Ε, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ε, πώς είναι δυνατόν να προκρίνεται μια λύση χωρίς να έχει προηγηθεί μια ενδελεχής μελέτη επιπτώσεων και πιο συγκεκριμένα, επειδή το είπατε και πριν στην απάντησή σας προς την κυρία Μακάρθη, κάνατε λόγο για τον κίνδυνο να υπάρξει πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρώπη από την εφαρμογή ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και στην ανακοίνωση της Επιτροπής ε, κάνετε αναφορά στην πιθανότητα διαφυγών κερδών στην περίπτωση που εφαρμοστεί φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πώς τεκμηριώνεται ότι θα έχουμε πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα ή κίνδυνο για διαφυγόντα κέρδη στην περίπτωση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ενώ δεν θα έχουμε τέτοιο κίνδυνο στην περίπτωση που προχωρήσουμε σε ένα φόρο επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος, σας ευχαριστώ πολύ. Θα πω, άλλωστε έχουμε συζητήσει, έχω συζητήσει και μαζί σας το θέμα αυτό στη συνάντησή μας. Μέσα στο τρέχον έτος έχουμε συντάξει μια αρκετά λεπτομερή ανάλυση της φορολογίας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όχι μόνο εμείς βέβαια γνωρίζουμε και την εργασία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου επίσης έχει κάνει λεπτομερή ανάλυση της φορολογίας του χρηματοπιστωτικού τομέα και όπου επίσης συμπεραίνει ότι ο φόρος επί των συναλλαγών έχει θετικές αλλά έχει και αρνητικές πλευρές και προτείνει το Ταμείο να εξεταστεί και το ενδεχόμενο επιβολής φόρου επί των δραστηριοτήτων ως εναλλακτική επιλογή. Αυτές οι αναλύσεις μας έχουν οδηγήσει σε ένα πολιτικό προσανατολισμό που λάβαμε ήδη τον Οκτώβριο και να πούμε ότι ναι, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα ήταν καλή ιδέα στο παγκόσμιο επίπεδο αλλά στο παρόν στάδιο δεν είχαμε σαφείς ενδείξεις ότι ο φόρος επί των συναλλαγών δεν θα οδηγήσει σε μετακίνηση αλλού των συναλλαγών και να λάβει υπόψη πόσο εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα μάλιστα που είναι μηχανο, μηχανογραφημένα πλέον όλα τα συστήματα του trading, να μετακινηθούν επομένως οι συναλλαγές σε άλλες αγορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Είναι βέβαια υψηλός ο κίνδυνος αυτός. Και όταν απάντησα στην πρώτη ερώτηση είπα ότι είναι επίσης σαφές ότι στην διαδικασία της Σύνταξη μελέτης επιπτώσεων που θα κάνουμε στους επόμενους μήνες, θα αξιολογήσουμε και άλλες εναλλακτικέ επιλογές. Φόρος επί των δραστηριοτήτων, φόρος επί των συναλλαγών, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στο παγκόσμιο επίπεδο, χρήση διαφορετικής ευρύτητας της φορολογικής βάσης. Πολλά θα εξαρτηθούν επίσης όπου το πόσο ευρεία είναι η φορολογική βάση και όσο πιο στενή είναι η φορολογική βάση τόσο πιο ε, άνισες καταστάσεις ε, δημιουργούμε ανάμεσα στους διάφορους μηχανισμούς φορολόγησης και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όλα αυτά τα θέματα θα αναλυθούν στην διάρκεια της ε, σύνταξη μελέτης επιπτώσεων και μετά θα αποκρισταλώσουμε απόψεις σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε με την φορολόγηση του τομέα αυτού. Το σύστημα φορολογίας μας ως τέτοιο ασφαλώς έχει κάποια αδύναμα σημεία σε ό,τι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα που είναι απειλαγμένος ΦΠΑ και θεωρούμε ότι θα ήταν ένα καλό μέσο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό ένας φόρος επί των συναλλαγών. Και σε ό,τι αφορά την μετακίνηση, η μεταφορά ολόκληρων επιχειρήσεων είναι πολύ πιο δύσκολη από τη μεταφορά απλώς των συναλλαγών. Και αυτό είναι ένα από τα κύρια επιχείρηματά μας. ότι δηλαδή ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων δεν συνεπάγεται τους ίδιους κινδύνους που ενδέχεται να συνεπάγεται ο φόρος επί των συναλλαγών. Λάβαμε τον πολιτικό αυτό προσανατολισμό βασισμένη στην ανάλυση που είχαμε μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ο Ούντο. Κύριε Επίτροπε, θα σας πω με καθόλου διπλωματικό τρόπο ότι δεν έχω την αίσθηση ότι διαβάζουμε τις ίδιες εφημερίδες με τον πρωινό μας καφέ όταν θέλουμε να συζητήσουμε πολιτικά θέματα. Μιλούμε τώρα πια για εντελώς τεράστια ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες για να στηρίξουν ένα σάπιο τραπεζικό σύστημα. 30-40% του ΑΕΠ μας για να σώσουμε τις τράπεζες. Τώρα μιλούμε για διαρκείς μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσεων. Τώρα στην Ιρλανδία πρέπει να αφαιρέσουμε 10 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό τους για να στηριχτεί η χώρα. Επομένως υπάρχει τεράστια πίεση στις κοινωνίες. Και μπροστά μας βλέπουμε μια κομισιόν η οποία εξακολουθεί να σέρνει τα πόδια της σε ό,τι αφορά το θέμα των εσόδων. Των εσόδων και κυρίως στους τομείς εκείνους όπου υπήρξαν κέρδη από κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Και όπου αυτοί που απεκόμισαν κέρδη από κερδοσκοπικές δραστηριότητες πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να συμβάλλουν. Είναι αρκετά δύσκολη και ε, δραματική κατάσταση ώστε να μην χρειάζεται να σας δώσω και άλλα πιο δραματικά παραδείγματα. Το Κοινοβούλιο ζήτησε μια μελέτη επιπτώσεων για την Ευρώπη, όχι παγκόσμια, για τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μας λέτε τώρα ότι ε, σας φαίνεται καλύτερος ο φόρος των δραστηριοτήτων. Ε, δηλαδή αυτοί οι φόροι που θα επιβληθούν σε αυτούς που κάνουν απλώς ενέργειες με τις τράπεζες, πράξεις με τις τράπεζες και όχι εκεί όπου υπήρξαν τα κερδοσκοπικά κέρδη. Δύσκολα μπορώ να κατανοήσω την επιχειρηματολογία σας. Άλλωστε τι αξία έχει ο λόγος σας όταν υποσχεθήκατε δηλαδή, αφού σας το ζήτησαν κιόλας, να ε, μελετήσετε τον φόρο επί των συναλλαγών. Θα πάρετε τα παλιά σας συμπεράσματα και απλώς θα τα αντιγράψετε στη νέα σας έκθεση ή υπάρχουν νέες μελέτες, νέες αναλύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να, υπάρχουν, για να έχουμε νέα, φρέσκια, ξεκάθαρη επιστημονική θεμελίωση και εν πάση περιπτώσει έχω λίγο κουραστεί με αυτό το κρυφτούλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά που μας λέτε εδώ είναι και οι αντιλήψεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνεί και αυτός ότι η αδράνεια στο θέμα της ε, φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι η σωστή στάση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν ναι, πρέπει να το συζητήσουμε. Εάν όχι, πάλι πρέπει να το συζητήσουμε. Ο Επίτροπος. Θα ήθελα να τονίσω ότι τους τελευταίους μήνες εργαστήκαμε, κάναμε τεράστιο έργο στον τομέα αυτό. Είμαι υποχρεωμένος να απορρίψω τα παράπονά σας ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κάνει τη δουλειά της. Κάνουμε πολλά πράγματα. Αναλύουμε την κατάσταση. Είναι εύκολο βέβαια να πει κανείς ας επιβάλλουμε τον ένα ή τον άλλο φόρο. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να αξιολογήσω ποιες θα είναι οι συνέπειες ή ασδήποτε τέτοιας αποφάσεως. Διότι εάν οι κίνδυνοι που διαβλέπουμε αυτή τη στιγμή υλοποιηθούν και οι συναλλαγές μετακινηθούν σε άλλες αγορές, τότε τα έσοδα που θα αναμέναμε από τον φόρο αυτό θα είναι πολύ χαμηλότερα από τις ε, προσδοκίες μας. Και τα ωφελήματα δεν πρόκειται, αυτά που αναμένουμε δηλαδή, να υλοποιηθούν. Άρα υποχρεώμεθα να αναλύσουμε την κατάσταση και τις συνέπειες μια ενδεχόμενη απόφαση και μάλιστα ιδιαίτερα προσεκτικά. Έχουμε εμπειρίε μέχρι τώρα και οι εμπειρίε που έχουμε δεν δείχνουν ότι ο φόρος αυτός στις χώρες εκείνες όπου έγινε προσπάθεια να επιβληθεί λειτουργήσε καλά. Γνωρίζουμε ότι η Σουηδία προσπάθησε να επιβάλλει το 1992 και οι συναλλαγές μετακινήθηκαν από τη Σουηδία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε και την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάποιος διακόπτει χωρίς μικρόφωνο. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να συζητηθεί το θέμα και με τις ίδιες τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, πώς λειτουργεί δηλαδή το σύστημα και τι αποδίδει. Και πρέπει να κατανοήσουμε επίσης πρέπει να συζητήσουμε και τις τεχνικές λεπτομέρειες. Ποια θα είναι η φορολογική βάση, πιο ε, ακριβώς τι, ποια ακριβώς δράση ή πράξη θα φορολογείται. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρά θέματα αυτά και η Κομισιόν τα εξετάζει αυτά πολύ σοβαρά και θα υποβάλουμε μια ανάλυση πραγματικά σε βάθος των ενδεχόμενων λύσεων. Και βέβαια και πρέπει να αξιολογήσουμε και άλλες προτάσεις ή και αποφάσεις στον τομέα αυτό. Καθώς επίσης και την αξιολόγηση του σωρευτικού αποτελέσματος των μέτρων που θα ληφθούν. Γνωρίζουμε ότι η Βασιλεία 3 θα επιβάλλει ορισμένες απαιτήσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα Έχουμε και το τέλος επί των τραπεζών που έχει συμφωνηθεί, εφόσον συμφωνηθεί μάλλον από τις χώρες μέλη, θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για τα Bank Resolution Funds. Έχουμε τον φόρο επί των συναλλαγών των φόρων επί των δραστηριοτήτων. Έχουμε τέλος πάντων μια παρέτα μέσων που πρέπει να αναλύσουμε και όπως είπα και το σωρευτικό αποτέλεσμα της χρήσης όλων αυτών των μέσων είναι Προ το συμφέρον μα, ο χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστικό παγκοσμίω. Να χρηματοδοτεί τι επιχειρήσει μα, και να έχει και το τμήμα που του αναλογεί στη συνολική ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το ερώτημά μου αφορά το CCTP, τα Ταμεία Εξυγίανσης Τραπεζών και δεν ξέρω κατά πόσο θα, μπορούσαν να, ε, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την φοροδιαφυγή, τη διασυνοριακή φοροδιαφυγή. Ε, μέσα στα πλαίσια του ε, διευρωπαϊκού εμπορίου. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως αυτή η φορολόγηση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών οδηγεί στους στόχους αυτούς. Χαίρομαι διότι συμφώνησαν μαζί μου πολλοί ε, βουλευτές και στο Κοινοβούλιο έγινε ένα λεπτομεριακό σεμινάριο σε σχέση με τις ομαδοποιήσεις φορολογήσεων προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε και είχαμε και πολλές ε, περίπλοκες ερωτήσεις. Δεν ξέρουμε πώς γίνεται η τιμολόγηση μεταφορών ε, στο, στο εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων. Πώς ορίζουμε δηλαδή τα κέρδη τα οποία μετά θα φορολογηθούν. Μιλάμε λοιπόν για τον φόρο σε ένα ενοποιημένο επίπεδο. Γιατί μας ενδιαφέρουν οι διάφοροι παράγοντες. Θα πρέπει να δούμε κατά πώς θα γίνει κατακαιρματισμός ανάλογα με τα στοιχεία ενεργητικού, τη μισθοδοσία και ούτω καθεξής. Και μετά θα γίνει μια πολιτική συζήτηση για τον επιμερισμό των ε, εσόδων από τη φορολόγηση και ξέρουμε ότι πολλοί θα μετακινήσουν τα στοιχεία ενεργητικού για να φτάσουν σε μία διαιτησία του συστήματος και να ελαχιστοποιήσουν τους φόρους. Και υπάρχει και το θέμα του προαιρετικού χαρακτήρα, διότι λέμε ότι μία επιχείρηση μπορεί να συμφωνήσει να συμμετάσχει σε αυτό το φόρο ή όχι σε αυτό το κοινό ενοποιημένο εταιρικό φόρο, CCCT. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο ε, θα δεχτεί κανείς ένα προαιρετικό σύστημα. Τότε το κράτος μέλος θα πρέπει να έχει και τα δύο συστήματα. Άρα αυτό τι κάνει, αυξάνει τη γραφειοκρατία. Άρα, εάν είναι προαιρετικό ή αν δεν είναι, αυτό θα πρέπει να το ορίσετε ως προς τη μείωση της γραφειοκρατίας. Εμείς θέλουμε αναπτυξιακό ρυθμό για τις ε, επιχειρήσεις, μειώνοντας όμως τη γραφειοκρατία. Εάν μία ε, εταιρεία επιχείρηση δεχτεί αυτό το φόρο, τον κοινό ενοποιημένο εταιρικό φόρο, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το κάνει για νομικούς λόγους. Έχει γίνει και μία μελέτη αντικτύπου γιατί μπορεί να αυξήσει τη φορολόγηση κατά ένα 13%. Άρα αυτό δεν μειώνει ούτε καν τη γραφειοκρατία και αυξάνει και τη φορολόγηση. Άρα, Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι άλλες προτάσεις έχετε για να ενθαρρύνετε το διασυνοριακό εμπόριο απλουστεύοντας όμως το φόρο εκτός από το CCTB. Yeah, πολλά ζητήματα τα οποία εντάσσονται στη συζήτηση της Κομισιόν, γιατί όπως σας είπα, σε αυτή τη φάση προβαίνουμε σε μία μελέτη αντικτύπου και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τις διάφορες επιλογές να δούμε κατά πόσο έχουμε να κάνουμε με ένα προαιρετικό σύστημα. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία μεγάλη γκάμα επιλογής. Σε αυτή λοιπόν τη φάση θα δούμε ποια θα είναι η κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση, διότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις ως προς την ε, κοινή φορολόγηση, διτή φορολόγηση ή κοινή φορολόγηση. Και οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι υπέρ αυτής της ιδέας. Και μας ενδιαφέρει να δούμε τι θα αποφασίσει το Διευθυντήριο. Βεβαίως είναι πολύ δύσκολο αυτό το θέμα. Και θα γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα της ε, πρότασης για να μειώσουμε και το διοικητικό φόρτο. Και αυτό που αξίζει είναι να ε, εγγύψουμε σε αυτό το θέμα. Σε σχέση τώρα με άλλες εναλλακτικές, με ε, βάση το δικό μου χαρτοφυλάκιο ενδιαφερόμαστε για την μείωση εμποδίων στην εσωτερική αγορά και γι' αυτό ελπίζω να τα ε, καταφέρουμε και ως προς τις μελλοντικές ε, συζητήσεις για το ΦΠΑ, δηλαδή να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο και από τις εκτιμήσεις μας βλέπουμε ότι το σύστημα ΦΥΠΙΑ αποτελεί μεγάλο μέρος του διοικητικού φόρτου, εάν λάβουμε υπόψη και τις εξελίξεις των τελευταίων ετών. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα εξυγχρονισμένο σύστημα ΦΥΠΙΑ για να αντιμετωπίσουμε το διοικητικό φόρτο κατά των επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει και με τη διπλή φορολόγηση. Θα ε, προβώ σε μία ανακοίνωση στις αρχές του επόμενου έτους για να απλουστεύσουμε ε, τη ζωή των επιχειρήσεων. Το CCTB αυτός ο κοινός ενοποιημένη, κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις εταιρείες που στο εξής θα αναφέρουμε ως CCTB, νομίζω ότι ε, ενδεχομένως να βοηθά τις επιχειρήσεις, διότι έτσι μπορούν να προετοιμάσουν τις μελλοντικές τους εργασίες. Σαν Πολ. Κύριε Επίτροπε, από τη στιγμή που σας ακούω, θα ήθελα να σας πω ότι συμπάσχω μαζί σας, συμπάσχω βαθύτατα. Επαναλαμβάνει ο μιλητής ότι από τη στιγμή που σας ακούω θα ήθελα να σας πω ότι συμπάσχω μαζί σας. Γιατί συμπαθήν στα αρχαία ελληνικά σημαίνει συμπάσχω και όχι αυτό που νομίζουμε ε, ε, δηλαδή το συμπαθήν έχει την έννοια των ε, συλληπιτηρίων στην παρούσα περίπτωση. Δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Έχετε το δυσκολότερο χαρτοφυλάκιο διότι προσκρούεται στην αντίσταση των κρατών και στις πιέσεις των διαφόρων ομάδων πίεσης που προωθούν ένα περίπλοκο σύστημα φορολόγησης. Θα ήθελα να ε, επαναλάβω την ερώτηση του Μαργκάγιο γιατί ε, πιστεύω ότι με την επανάληψη η επανάληψη είναι μήτυρ πάσης μαθήσεως. Αυτό το ακούμε από το 2004. Ένας από τους προκατόχους σας έλεγε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Τότε γιατί να ακούσουμε τον ε, πρόεδρο της ε, ΕΚΤ, εάν δεν μπορούμε να φτάσουμε σε μία ενοποιημένη βάση, τότε χάνουμε το χρόνο μας. Άρα αυτή είναι και η ερώτησή μου. Πότε θα έχουμε μία ενοποιημένη βάση και φιλικά θα ήθελα να σας πω ότι μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό το κοινοβούλιο για θέματα φορολόγησης. Δεν έχουμε ε, την, καταρχήν την αρμοδιότητα σε αυτό το θέμα, αλλά έχουμε μεγάλη πείρα. Γιατί τι ζητούν οι συμπολίτε μας, πού βρισκόμαστε ως προς την ε, φορολόγηση στην Ευρώπη. Βασιζόμαστε σε εσά και πάλι θα ήθελα να σας πω ότι συμπάσχω, μαζί σας βαθύτατα και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ενθαρρυντικά αυτά λόγια. Εγώ θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι φυσικός μου σύμμαχος στη δουλειά που κάνω και βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξω το Συμβούλιο σε κάποια απόφαση γιατί υπάρχουν και τα, οι κανόνες πλειοψηφίες και τα λοιπά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επηρεάσει ε, πολύ τις προσπάθειές μου, το Συμβούλιο, στη θέση που θα πάρει για τις προσπάθειές μου για τις αρμοδιότητες μου είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό επίσης οι ευρωβουλευτές να δρούν ε, έγκαιρα και στα κράτη-μέλη τους, στο εσωτερικό των μελών τους, για να προωθηθούν ορισμένα ζητήματα. Και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να αρχίσουν να κουβεντιάζουν αυτές τις ιδέες και να πιέσουν αν θέλετε τις κυβερνήσεις να επηρεάζουν τις κυβερνήσεις ε, στις προτάσεις τις οποίες ε, υποβάλλουν και πραγματικά Νομίζω ότι όταν φτάσουμε σε ένα σημείο κατά το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται και με τα εθνικά και με εμά, ε, τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Ε, ως προς την ε, φορολόγηση των επιχειρήσεων, θα ήθελα να σας πω ότι δεν πρόκειται για μια πρόταση που προστίθεται σε όλες τις άλλες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχει μία ρύθμιση των αγορών κατά αυτόν τον τρόπο. Και ως προς τις ε, χρηματοδοτικές δυνατότητες, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να την δείτε σοβαρά, όχι να τη δείτε σαν μία μεταξύ άλλων. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά την Ιρλανδία. Η φορολόγηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών. Η Ευρωζώνη όμως σήμερα πλήττεται από μεγάλες μακροοικονομικές ισορροπίες. Δεν πιστεύετε ότι στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης σε αυτό το βαθμολόγιο που θα ε, θέσουμε σε ισχύ δεν θα πρέπει να εισαγάγουμε και στοιχεία φορολόγησης, διότι βλέπουμε ότι στο Ιρλανδικό μοντέλο η στρατηγική των πολυεθνικών δεν μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας, δεν μπορεί να οδηγήσει στην άρδευση της οικονομίας δηλαδή σχηματικά. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε και συντελεστές φορολόγηση στο βαθμολόγιο αυτό μέσα στα πλαίσια της μακροοικονομικής εποπτείας. Δεύτερον, στα πλαίσια της παρούσας θητείας ασχοληθήκαμε με την φορολόγηση των αποταμιεύσεων και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα αυτόματο σύστημα πληροφόρησης με τους εταίρους. Πριν και από την κρίση μιλήσαμε για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Βεβαίως η κρίση επιδίνωσε τα πράγματα και ο πρόεδρος του Διευθυντηρίου σας μίλησε για την ανάγκη καταπολέμησης των φορολογικών παραδείσων. Εάν λοιπόν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα, δεν θα πρέπει να έχουμε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Δύο όμως κράτη-μέλη βασίζονται σε ένα σύστημα καταγγελιών και μαζί με την ε, Ελβετία έφτασαν ε, σε μια συμφωνία η οποία υποβαθμίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με την Ελβετία. Και έτσι ένα κράτος μέλος έχει ανακτήσει 30 δις ευρώ ε, κατά όμως της αλληλεγγύης, της ενδοκινοτικής αλληλεγγύης, στις διαπραγματεύσεις με την Ελβετία. Πιστεύετε ότι έτσι καταπολεμούμε τους φορολογικούς παραδείσους τη στιγμή που τα κράτη-μέλη πρέπει να ανακτήσουν έσοδα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουν να εφαρμόσουν και το πρόγραμμα λιτότητας. Ε, εγώ θα κάνω πρώτα μία σύντομη παρατήρηση για την φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα που στο πρόγραμμα της Κομισιόν είναι μια σημαντική στρατηγική πρωτοβουλία την οποία επεξεργαζόμαστε και έχω αναλάβει δέσμευση να οδηγήσω σε πέρας την προσπάθεια αυτή. Σε ό,τι αφορά την οικονομική διαχείριση και τα θέματα φορολόγησης, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι στο παρελθόν την πιο πολύ προσοχή μας σχετικά με τις διαδικασίες ε, υπερβολικού χρέους στις χώρες μέλη είχαν σχέση με το τμήμα των δαπανών, των εξόδων και λιγότερο των εσόδων όταν αξιολογούσαμε την κατάσταση μιας χώρας μέλους. Γι' αυτό τώρα εγώ επεξεργάζομαι τώρα αυτό το κόνσεπτ, αυτή την έννοια της ποιότητας των εσόδων που θα είναι και μέρος των μηχανισμών που θα έχουμε στη διάθεσή μας για να αξιολογήσουμε το τμήμα εσόδων, την πλευρά των εσόδων των χωρών μελών, την μακροοικονομική τους κατάσταση, καθώς και τις προβλέψεις για τις μελλοντικέ εξελίξεις, μακροοικονομικά δηλαδή, των χωρών μελών. Νομίζω ότι πρέπει να εγκύψουμε στο θέμα αυτό και πρέπει να αναπτύξουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς για να το υλοποιήσουμε. Είναι πράγματι μια εργασία που προχωρεί. Για το θέμα των φορολογικών παραδείσων και του τρόπου αντιμετώπισης τους, είναι αληθές ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούμε την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως ένα μέσον που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε αμέσως το θέμα. Έχουμε τώρα και τα στάνταρτ του ΟΣΑ, που λέει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται κατόπιν και άλλες χώρες στον κόσμο που προχωρούν στην εφαρμογή των προδιαγραφών του ΟΟΣΑ. Πρόσφατα επισκέφθηκα το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο, που ενέκριναν πρόσφατα νομοθεσία, φέτος δηλαδή, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Εμείς εξακολουθούμε... Δεν έχει μικρόφωνο η υπηρέσεις. Ναι, απάντηση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα στο οποίο θα επανέλθω, αλλά στο διεθνές πλαίσιο, για παράδειγμα τον Απρίλιο περάσαμε την ανακοίνωση για τον φόρο και την ανάπτυξη και επίσης και στην ανακοίνωσή μας για την εμπορική πολιτική έχουμε βάλει ρήτρα περί φορολόγησης στις πολιτικές μας και όταν διαπραγματευόμαστε συμφωνίες με τρίτες χώρες θα διαπραγματευόμαστε και θέματα χρηστής οικονομικής διαχείρισης με τις χώρες αυτές. Άρρωστε βρισκόμαστε ήδη μέσα στα πλαίσια των ε, διαβουλεύσεων με τρίτες χώρες για τα θέματα αυτά. Και σε ό,τι αφορά το θέμα με την Ελβετία, είναι γεγονός ότι η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις με την χώρα αυτή και το υφιστάμενο πλαίσιο δεν απαγορεύει στις χώρες αυτές να προχωρήσουν στη σύναψη συμφωνιών αρκεί βέβαια να μην αντιβαίνουν αυτές οι συμφωνίες στους κανόνες που ήδη ισχύουν. Εγώ πιστεύω ότι και η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν και να προωθήσουν τις αρχές αυτές μέσα σε δύσκολες όντως διαπραγματεύσεις με την Ελβετία για τα θέματα αυτά. Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν είναι και τόσο απλές όπως μας λένε ορισμένες πηγές καμιά φορά. Και θα δούμε βέβαια και ποια θα είναι και η εκβασή τους των διαπραγματεύσεων αυτών. Ευχαριστώ. Εσείς, Σβέν. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που προσήλθατε και που προχωρείτε σε αυτή την όχι εύκολη συζήτηση για ένα θέμα βαρύ. Συμφωνώ με τον Ζαν Πολ ότι δηλαδή ε, θεωρούμε ότι εσείς βρίσκεστε σε δύσκολη θέση μέσα σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο επίσης είναι δύσκολο. Νομίζω πάντως ότι έχει αλλάξει η κατάσταση και δεν είμαι βέβαιος για το εάν πράγματι έχετε πλήρως ενσωματώσει την αλλαγή αυτή στην στρατηγική σας και στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε εδώ αλλά και στις προτάσεις που κάνετε. Εξετάζοντας την οικονομική διαχείριση, η διακυβέρνηση, ορισμένα πράγματα που εγκρίνονται τώρα ήταν λίγο πολύ αδιανόητα και πριν από λίγους μήνες. Γνωρίζω από τη Γερμανία την κατάσταση και ξέρω για ποιο πράγμα μιλώ. Η φορολόγηση των ε, ε, χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων θα ήταν αδιανόητη πριν από λίγο καιρό. Τώρα, χρειάζεται μια σταδιακή προσέγγιση, η οποία όμως δεν συμβαδίζει με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, όπου χώρες, οι χώρες μέλη έχουν τεράστια ελλείμματα και ταυτόχρονα υπάρχουν εισοδήματα τα οποία είτε είναι αφορολόγητα είτε είναι φορολογημένα με πολύ ελαφρούς συντελεστέ. Και όμως λέτε ότι δεν θέλετε ελάχιστους φορολογικούς συντελεστές ακόμα και για τα πιο ευκίνητα εισοδήματα. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η στάση δεν είναι προσαρμοσμένη στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν, κάνετε προτάσεις στου διάφορου τομεί, Προτάσεις όπως κάνουν οι άλλοι συναδελφοί σας, Όλοι Ρεν και Μισελ Μπαριέ για να πάτε στο Συμβούλιο και να έχετε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για πρώτη φορά οι συντονιστές εδώ στην ε, ε, Οικονομική Επιτροπή συμφώνησαν και υπέγραψαν ότι θα υποστηρίξουν ε, φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις του 25%, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο πριν από λίγο καιρό. Επίσης θα συμφωνήσω με πολλές από τις γνώμες που, εξέφρασαν οι συναδελφοί μου. Τώρα, για την ανταλλαγή πληροφοριών. Για το 2011, στον κατάλογο μέτρων δηλαδή, δεν το βρήκα αυτό και αυτό είναι κρίμα διότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει κατ' επανάληψη να θεσπιστεί. Θέλω να μάθω εάν πρόκειται να υποστηρίξετε τον συνάδελφό σας της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς για τα μέτρα αυτά. Και τέλος, απευθύνω έκκληση. Να ξεφύγετε από το όχι και το όχι προχωράμε προσεκτικά σε μια πιο θαραλέα ανάληψη δράσεως, ανάληψη των ε, ευθυνών σας, γνωρίζοντας ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζετε είναι δύσκολη. Αλλά οι υπερχρεωμένες χώρες που χρειάζονται υποστήριξη από τις κυβερνήσεις των εταίρων χωρών τους θα έχουν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να δεχθούν τέτοιες προτάσεις αν περάσει λίγος καιρός ακόμα. Ωραία λοιπόν. Θα φροντίσω να υποβάλω τις προτάσεις και στα τελευταίες ε, στα τελευταία συμβούλια ΕΚΟΦΗΝ σε κάθε συνεδρία, σύνοδο των Υπουργών Οικονομίας στα πλαίσια του ΕΚΟΦΗΝ το Συμβούλιο ε, συζητούσε θέματα φορολογίας και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πιστέψτε με, οι συζητήσεις αυτές δεν είναι εύκολες και τα κράτη-μέλη δεν ε, συμφωνούν για όλα υπάρχουν ε, σοβαρές διαστάσεις απόψεων ακόμη ε, και πρέπει να παρουσιάσουμε μια πολύ σαφή ανάλυση της κατάστασης, να περιγράψουμε Το ωφέλη που θα αποκομίσει κανείς από την αλλαγή της κατάστασης κτλ. Τώρα βέβαια οι εκθέσεις αναχώρα, όντως αυτό το θέμα βρίσκεται επιτάπητος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα είμαι στο στάδιο των δημοσίων διαβουλεύσεων για το ζήτημα. Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από τις διαβουλεύσεις και θα υποβάλουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας βεβαίως και το εξή. Είναι προφανές ότι οι ανεκθέσει ξεχωριστές αναχώρα θα βοηθήσουν όμως η φορολογία ότι ουσιαστικά το να δώσει κανεί στοιχεία για τη φορολογία και τη φορολογική κατάσταση ουσιαστικά είναι σαν να δίνει στοιχεία για επιχειρήσεις και λεπτομέρειες για επιχειρήσεις. Εκεί υπάρχει, ε, πρέπει να τα προσέξουμε αυτά τα πράγματα ε, αλλά είμαι σίγουρο ότι όταν υπάρξουν οι εκθέσεις αυτές αναχώρα θα είμαν τα πράγματα πιο ξεκάθαρα. Ε, Λοιπόν, τώρα έχουμε Φίλιπ Λαμπερθ. Προσθέθηκαν ένα-δυο ομιλητέ. Φιλίπ, ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το 19ο αιώνα όταν ε, πρωτοακούγονταν οι έννοιε τη ε, κοινωνική ασφάλισης κτλ., υπήρχαν φωνές που λέγανε stop, stop, stop, αυτό θα σκοτώσει την κοινωνία, μην το κάνετε. Την οικονομία, με συγχωρείτε. Μετά ήρθε η έννοια του φόρου που στέμενες αξίες και πάρα πολύ φωνάζανε ότι μην το κάνετε θα σκοτώσετε την οικονομία. Ορίστε, έχουμε ΦΠΑ, έχουμε κοινωνική ασφάλιση, δεν έχει σκοτωθεί η οικονομία. Και τώρα στον 20ο ε, αιώνα φωνάζουν, φωνα, 21ο αιώνα φωνάζουν ε, μην εφαρμόστε το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών διότι μπορεί να μην σκοτώσει αυτό στην οικονομία αλλά θα σκοτώσει τις συναλλαγές. Δεν είμαι σίγουρος κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, κυρία Πρόεδρε. Είναι... <coughs> Είναι σημαντικό, δεν λέω να σωθούν οι τράπεζες αλλά χωρίς συμβολή των τραπεζών οι κυβερνήσει είναι σημαντικό να κάνουν οικονομίες αλλά πρέπει να το κάνουν τόσο γρήγορα η έννοια αυτή του κατεπήγοντος που διέπει αυτού του είδους τις προσπάθειες από πού προήρχε έγινε καμιά ανάλυση του σωρευτικού αποτελέσματος αυτών των μέτρων έγινε ανάλυση του αντικτύπου στην οικονομία αντίκτυπος των, των επιγόντων αυτών και ε, βίων και τα γρήγορων μέτρων στην οικονομία. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν το σωρευτικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια κάποια ανάλυση. Λοιπόν, σιγά σιγά, γιατί να βιαζόμαστε. Κάνουμε πρώτα τις μελέτες αυτές. Μας λέτε επίσης ότι υπάρχει ανταγωνισμό στο, στη φορολογία, αγώνα στη φορολογία. Ε, αν θέλετε, ε, δείτε, οι κυβερνήσεις δεν είναι όλες καλές, δεν τους κάνει κακό και λίγο να προσέξουν τη φορολογία. Από εκεί και πέρα εκείνο που βλέπουμε δείτε τι συμβαίνει γύρω μας δείτε τι συμβαίνει από κάποιους βασικούς φορείς της οικονομίας είναι And it's not you personally, είναι αδιφάγοι κάποιοι φορείς εμείς τι κάνουμε Για, γιατί εκεί δεν είμαστε γρήγοροι Επίτροπος για να απαντήσω εν συντομία τι να πω, εσείς ο ίδιος θα μας επικρίνατε εάν είχαμε υποβάλει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για οδηγίες στο φορολογικό τομέα δίχως να κάνουμε λεπτομερείς αναλύσεις. Το θέμα δεν είναι μια, προ, μια απόφαση η οποία επηρεάζει το ένα ή το άλλο κράτος μέλος. Επηρεάζει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι απαραίτητες οι αναλύσεις αντικτύπου εδώ. Και πρέπει να γίνει μια μελέτη λοιπόν των, επιδρα... των επιπτώσεων σε βάθος. Uh, δεν είναι γεγονός ότι δεν είναι γεγονός ότι διάφορες κυβερνήσεις μοναχά ασχολούνται με την ε, ε, πλευρά ή επιβάλλουμε να ασχολούνται με την πλευρά των δαπανών. Πάρτε την Ελλάδα, πάρτε την Ιρλανδία και η μεριά των εσόδων ε, μελετάται και πολλά μέτρα εφαρμόστηκαν και στην ε, Ιρλανδία και σίγουρα στην Ελλάδα για τον επηρεασμό των εσόδων. Λοιπόν δεν είναι αλήθεια ότι όλα τα μέτρα ε, που παίρνονται από τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν ορισμένα αυτά τα μέτρα βρίσκονται στην πλευρά των δαπανών. Η Σόφη. ένα ίσονο σημασία, ένα μικρούλι ερώτημα, εν πάση περιπτώσει, για το ΦΠΑ. Έστειλα γραπτή την ερώτησή μου, μου στείλατε μια απάντηση, δεν με ικανοποίησε. Τώρα, γιατί άμα ε, αγοράσω την καλύβα του Παρπαθωμά ε, σε paperback, πληρώνω λιγότερο φόρο από ότι για τα ηλεκτρονικά βιβλία και το audio, τα audiobooks παραδείγματο χάρη. Προωθούμε δηλαδή το παραδοσιακό βιβλίο, το χάρτινο βιβλίο σε αντίθεση με κάποια καινοτόμα προϊόντα. Νομίζω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Επίτροπος, ξέρετε το δίχως άλλο ότι έγινε το 2009 μια μεγάλη συζήτηση για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή του ΦΠΑ για ορισμένους κλάδους. Συζητήθηκε στο Συμβούλιο αυτό και επετέφθη συμφωνία εκεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης τότε ήμουνα υπουργό οικονομικών της χώρας μου σε εκείνη και τη συζήτηση λοιπόν έγινε λόγος για μειωμένους φορολο... συντελεστές ΦΠΑ για τα βιβλία στο διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά βιβλία και τα audiobooks. Όμως η πρόταση αυτή δεν υποστηρίχθηκε από τα κράτη-μέλη. Δεν συμφώνησαν τα κράτη-μέλη να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ για αυτά τα προϊόντα. Η συζήτηση πάντως γενικότερα των μεωμένων συντελεστών ΦΠΑ είναι ευρύτερη και αύριο θα συζητήσουμε όταν θα, συζητήσουμε, θα συζητήσουμε για το μέλλον του ΦΠΑ και θα γίνει ακριβώς κουβέντα για όλα αυτά, για τις απαλλαγές, για τις εξαιρέσεις, για τις, τους μειωμένους συντελεστές. Εγώ προσωπικά πιστεύω πως θα ήταν καλή ιδέα να εξισωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ. Βέβαια, Το ερώτημα είναι πού θα εξισωθούν οι συντελεστές στο ψηλό επίπεδο ή στο μειωμένο επίπεδο. Τέλος πάντων, αυτό θα είναι το αντικείμενο της συζήτησης που βασίζεται και στην πράσινη βίβλο. Αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μπορεί να επιτευχθεί ομοφωνία για οποιουσδήποτε μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ διότι η απόφαση που πέρθηκε πέρσι ε, στη συναπόφαση που πάρθηκε οχτώ κράτη-μέλη έκαναν ε, δηλώσεις που, στις οποίες λένε ότι είναι κατά της γενικότερης διεύρυνσης των μειωμένων συντελεστών. Όμως στη διάρκεια της συζήτησης για την Πράσινη Βίβλο σίγουρα θα συζητηθεί το θέμα αυτό και έτσι θα ακούσουμε και τη γνώμη των ενδιαφερομένων. Ρόντι. Ε, θα, θα σας κάνω μια ερώτηση η οποία δεν απέχει και πολύ από αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τάσεις των φορολογικών συστημάτων στο 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει σημαντικές διαφορές ως προς την ε, άντληση συνολικών φορολογικών εσόδων. Θα ήθελα να ρωτήσω αν στο πλαίσιο του συντονισμού των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών και της ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς θα μπορούσε ε, να συνεισφέρει και η άμβληση των διαπιστωμένων διαφορών μεταξύ των εθνικών φορολογικών συστημάτων τόσο ως τη φορολογική πολιτική όσο και ως προς τα κοινά κριτήρια στο πλαίσιο μιας καλής φορολογικής διακυβέρνησης. Και αν ναι, πώς θεωρεί η Επιτροπή ότι θα επιτευχθεί αυτή η σύγκληση ε, που θα συμβάλλει και στην επίτευξη ενός δίκαιου φορολογικού ανταγωνισμού. Ευχαριστώ πολύ. Uh, well, Ένας από τους στόχους της Πράσινης Βίβλου για τον ΦΠΑ θα είναι με ποιον τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η σωστή η λειτουργία της ενίας αγοράς με μειωμένους συντελεστές, με εξαιρέσεις από ΦΠΑ, με συστήματα εκπτώσεων πού θα πρέπει να επιβάλλεται ο φόρος στον, ε, στη χώρα ε, της προσφοράς ή ε, της αποδόσεως και ούτε καθεξής. Όλα αυτά θα συζητηθούν και στη βάση της συζητήσεως αυτής θα καταλήξουμε, θα αναπτύξουμε μια νέα στρατηγική ΦΠΑ για τα επόμενα χρόνια. Και σε άλλους τομείς μέτρα όπου εφαρμόζουμε σχετίζονται με τον καλύτερο συντονισμό των φορολογικών συστημάτων με πρωτοβουλίες κατά της διπλής φορολογήσεως που θα υποβάλουμε και που θα αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό με πακέτα εξοικονομήσεων για καλύτερη διαχείριση της ε, καταστάσεως στην ενιαία αγορά. Όλα αυτά εντάσσονται σε αυτή τη συζήτηση. την οποία διεξάγουμε τώρα σχετικά με την ποιότητα των εσόδων. Και αυτή η συζήτηση λοιπόν άπτεται μιας προσπάθειας καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών για φορολογικά θέματα. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να λησμονούμε τα θέματα κυριαρχίας των χωρών μελών, θέματα επικουρικότητας, γιατί οι χώρες μέλη επιθυμούν να διατηρήσουν το δικαίωμα να καθιερώνουν τα φορολογικά του συστήματα ανταποκρινόμενα στις ιδιαίτερες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστώ. Ο Γκέι, μάλλον. Γκέι Μίτσελ. Η προσαρμογή στην Ιρλανδία σήμερα θα είναι 6 δισεκατομμύρια ευρώ που θα ισοδυναμούσε με 60-70 δισεκατομμύρια ευρώ για τον Βρετανικό προϋπολογισμό, αν δηλαδή ήταν σε μετά του Βρετανικού προϋπολογισμού. Τα πάθη και τα δεινά των Ιρλανδών θα είναι βαρύτατα και με τα φορολογικά μέτρα. Υπό τις περιστάσεις αυτές είναι σημαντικό οι Γερμανοί και άλλοι φίλοι μας να δουν τι ακριβώς ε, σημαίνουν αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια μικρή χώρα όπως η Ιρλανδία περνά από ε, δύσκολες περιστάσεις τώρα, αλλά τι θα γίνει αν μια χώρα όπως η Πολωνία, για παράδειγμα, περάσει από τα ίδια. Κάποιος είπε ότι οι συντονιστές έχουν συμφωνήσει και υπογράψει να αυξηθεί ο φόρος του 25%. Δεν έπραξαν τέτοιο πράγμα οι συντονιστές. Όταν έθεσα το θέμα, μας είπε ο συντονιστής του Λαϊκού Κόμματος ότι υπέγραψε σε προσωπική βάση. Δεν έχει γίνει σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα γι' αυτό δεν πρόκειται να δεχθούμε να μας πιέσουν οι συντονιστές. Οι συντονιστές και στην παρούσα επιτροπή δεν έχουν παραπάνω από μία ψήφο όπως όλα τα άλλα μέλη. Γίνονται πράγματα εδώ τα οποία έχουν αναστατώσει πολύ τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Συζήτηση και συμφωνία είναι ο μόνος τρόπος με τον, με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ δεν ήμουν παρόν σε όλα σας τα σχόλια προηγουμένως. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα. Πολλοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονε θεωρούν πολλές από, την, πολλές από τις αλλοδαπές που είχαν έρθει στην Ιρλανδία μέχρι τώρα ήταν αμερικανικές και δεν πρόκειται τώρα να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάνε στην Ελβετία. Και εάν χρειάζεται μια διακυβερνητική διάσκεψη για να αλλάξουν τα πράγματα, ας γίνει αυτό τότε. Στο μεταξύ όμως, αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο που έχετε και είναι δύσκολο το έργο σας, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για αυτά τα πράγματα. Θα επιβάλλουμε φόρο ε, στα κέρδη των επιχειρήσεων. Η χώρα μου έχει πολλές μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν ε, γίνει incorporated ακόμα. Είναι πολύ ευαίσθητο ο τομέα λοιπόν αυτό και χρειάζεται προσεκτική αντιμετώπιση και πολλά λέγονται για του συντελεστέ του εταιρικού φόρου. Πολλά από αυτά δεν είναι ωραία, είναι άσχημα. Πολλοί λένε για τα όσα εισφέρουν οι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μη σμωρούν και τι συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στι ε, χώρε μέλη. Και κυρίω σε περιπτώσει όπου υφίσταται τα πάνδυνα οι ευρωπαϊκές ε, χώρες. Επανέρχομαι σε κάτι που είπε ένας συναδελφός μου για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Νομίζω είναι ένας τομέας όπου μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια να προχωρήσετε μαζί με τις χώρες μέλη. Υπάρχει μια περίοδος όπου αξίζει τώρα να συζητηθούν και να προωθούν νέες ιδέες τόσο, τώρα που έβλαψαν τόσο πολύ οι χρηματοπιστωτικές αγορές της χώρας. Μέχρι τώρα ρυθμιζόταν η χώρα μου από τον ιδιωτικό τομέα, από τις αγορές και από, τις, ε, από τους οίκους αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Αυτοί ρυθμίζαν και τον δημόσιο τομέα μέχρι τώρα. Τουλάχιστον τώρα ο, ο δημόσιος τομέας ρυθμίζεται από τον δημόσιο τομέα. Αλλά πρέπει τώρα να ε, συζητηθεί περισσότερο ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Κύριε Επιτροπέ, αυτό, αυτή είναι η γνώμη μου. Η Ιρλανδική κατάσταση βέβαια έχει επισύρει την προσοχή μας. Χθες όταν κάναμε την προπαρασκευαστική συνάντηση για τον ε, νομισματικό διάλογο τέθηκαν θέματα όπως της διαχείρισης και αντιμετώπισης της κρίσης και υπάρχουν πολλοί άλλοι φόροι εκτός από τον εταιρικό φόρο που συζητήθηκαν. Για παράδειγμα, παρενόησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να αντιμετωπιστεί η κρίση με τον φόρο επί της ακίνητης περιουσίας στην ε, ε, Ιρλανδία. Τώρα, βέβαια τα ρυθμίζουν αυτά. Μου φαίνεται σαφές ότι χρειάζεται περισσότερες, χρειάζονται περισσότερες προφορίες από τις ίδιες τις χώρες μέλη σε ό,τι αφορά την ανάλυση των φορολογικών, των τους βάσεων και πώς μπορούν να τα αποκριθούν σε αυτές τις ε, καταστάσεις εντάσσεως. Και χωρίς να αλλάξουμε τις συνθήκες θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε αυτό. Δεν μου φαίνεται να ε, είναι επικίνδυνο να συλλεχθούν οι πληροφορίες αυτές. Βέβαια πήρα ε, αφορμή από την ερώτηση του Γκάι, αλλά νομίζω ότι είναι περίπου στην ίδια, στο ίδιο μήκος Συμφωνώ μαζί σας ότι για να γίνει η αξιολόγηση της ποιότητας των εσόδων μιας χώρας μέλους θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις κατάλληλες πληροφορίες για το φορολογικό σύστημα στην συγκεκριμένη χώρα μέλος και οι πληροφορίες αυτές για τα φορολογικά συστήματα είναι και κλειδί για την σωστή αξιολόγηση της ποιότητας των εσόδων. Και πρέπει να βρούμε τρόπους, βέβαια ήδη συλλέγουμε πλήθος πληροφοριών από τις χώρες μέλη σε ό,τι αφορά τα φορολογικά του συστήματα Ορισμένες φορές αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι ορισμένες λεπτομέρειες των συστημάτων που είναι σημαντικές σε κάποια χρονικά διαστήματα δεν είναι πολύ καλά γνωστές. Χρειάζεται βελτίωση λοιπόν στην κατάσταση αυτή και στην βάση αυτή να εργαστούμε πάνω σε αυτή την έννοια της ποιότητας των εισόδων. και σε ό,τι αφορά τον ε, φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεν έχω περισσότερα να πω, εκτός από αυτά που είπα ήδη στη διάρκεια της συναντήσεως. Νομίζω προσωπικά ότι εάν χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, και στη συνεργασία μας, στην παγκόσμια συνεργασία μας, στα G, 20 Θα επιτύχουμε πρόοδο. Η Γαλλία έχει αναλάβει την προεδρία του G20 και θα συνεχίσουμε να προωθούμε την προσπάθεια αυτή και παγκόσμια τροφοδοτώντας την συζήτηση και με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και πορίσματα των αναλύσεων μας και της μελέτης επιπτώσεων. Όταν συζητούμε με τους διεθνείς εταίρους μας το θέμα αυτό και βέβαια είναι σημαντικό να συζητείτε όχι μόνο η φορολογία γενικά αλλά και οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες. της φορολόγησης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και γι' αυτό βασιζόμαστε και τόσο πολύ στη μελέτη επιπτώσεων. Ευχαριστώ. Ποιο ρολόι άραγε τα λέει σωστά. Μια τελευταία ερώτηση από τον ε, Ζωζέ. Ευχαριστώ. Στις ε, πρόσφατες παρεμβάσεις έγινε λόγος για τους τύπους ε, φορολόγησης μέσα στα πλαίσια της ενοποιημένης φορολογικής ε, βάσης. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο, ο πραγματικός αθέμητος ανταγωνισμός, ο οποίος μπορεί να ανακύψει από την υπέρμετρη φορολόγηση. Δεν μπορούμε δηλαδή το θέμα να το δούμε μεμονωμένα. και πιστεύω ότι ο, φόρος, ο εταιρικός φόρος ή φόρος ε, των επιχειρήσεων αφορά μία προστιθέμενη φορολόγηση, η οποία τουλάχιστον λειτουργεί ισορρευτικά ή προσθετικά. Πιστεύετε σε αυτή τη λογική ή όχι. Uh, uh, Σε σχέση με την φορολόγηση χρηματοοικονομικών ε, δραστηριοτήτων, πρόκειται για έναν φόρο που λειτουργεί ε, προσθετικά. Αποτελεί δηλαδή προσθέμενη αξία ως προς τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και ένα από τα ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία μελέτης αντικτύπου αυτού του φόρου είναι πώς να σχεδιάσουμε τον ίδιο το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δηλαδή, δεν πρέπει να περιορίσουμε τον αντίκτυπό του στους καταναλωτές ή τους πελάτες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να λειτουργήσει ένας φόρος χρηματοοικονομικής δραστηριότητας. Αυτό είναι ένα θέμα περιορισμένης μεταφοράς του φόρου στους καταναλωτές. Και αυτός είναι και ένας από τους στόχους ε, ε, υπολογισμού αυτού του φόρου, σχεδιασμού αυτού του φόρου. Ως προς τους ε, ε, δείκτες του εταιρικού φόρου, του συντελεστές του χρηματοοικονομικού αυτού φόρου, Αυτό θα το δούμε μέσα στα πλαίσια του CCTB. Και στόχος είναι να δημιουργηθεί διαφάνεια στο σύστημα. για να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος των ονομαστικών συντελεστών φορολόγησης έναντι των πραγματικών συντελεστών φορολόγησης. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που αν ε, συμφωνηθεί θα δημιουργήσει μια πιο σαφή κατάσταση στην ε, χρηματοπιστωτική αγορά ως προς την δραστηριότητα επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του CCCTB. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Θα σας ξαναδούμε σύντομα, δεν ξέρω πότε βεβαίως. Αλλά όπως και να έχει, θα ξανασυναντηθούμε και θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, ανακοινώσεις και προτάσεις της Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζω να δεχτείτε ορισμένες από τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοδομητική αυτή συζήτηση, λέει ο Επίτροπος. Και βεβαίως το Κοινοβούλιο είναι ο φυσικός σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την εργασία του επιφορολογικών ζήτημάτων. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσβατο αυτό το θέμα, αλλά προσμένουμε τη μελλοντική μας συνεργασία. Στην μελλοντική μας συνεργασία. Χαίρετε.